Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση, διότι αναμένουμε τον Ισπανό Γενικό Γραμματέα σύντομα να ξεμπερδέψουμε τα δικά μας, αν έχει την καρσία να καθίσετε, πάμε τον άκρο στο άλλο. Από, την, τερά, από την ωραία κυκλική μας αίθουσα, σε αυτή την τεράστια αίθουσα, αν το ακροατήριο ή θεατές επιθυμούν να μετακινηθούν προς το πρόστιο μέρος της αιθούσης, καλούνται να το κάνουν. Γίνεται πιο οικογενειακή ατμόσφαιρα έτσι. Στην ομίχλη του βάθους, μόλις που σας διακρίνουμε, λοιπόν, άμα θέλετε, λάτε πιο κοντά. Λοιπόν, το απόγευμα έχουμε ε, πολλά σημεία και πολλά εναρκτήρια σχόλια έχουμε κάνει. Πρέπει να είμαι αυστηρό με το χρόνο. Θα αποθαρρύνω μακροσκελείς παρεμβάσεις γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ξεκινάμε όμως τη διαδικασία συζητήσεως πολλών νέων θεμάτων. Εστέ υπομονετική απέναντί μου, διότι θέλω να τα καλύψουμε όλα απόψε και να μην αφήσουμε κρεμότηση για την επόμενη φορά που θα γίνει ουσιαστική συζήτηση. Πρώτο σημείο προς συζήτηση επίσημη έγκριση από την Επιτροπή ενός θέματος που συζήτησαν οι συντονιστές την Τρίτη και εξετάστηκε αρκετά λεπτομερώς η, μια, λόγω της ε, υιοθέτηση της ε, συνθήκης της Αβώνας προκύπτει το εξής. Μας έστειλε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να εξετάσουν όλων τους, τους καταλόγους των εκκρεμών διαδικασιών για να δουν κατά πόσο είναι πλήρης κατά πόσο στήν είναι η νομική βάση και ενδεχόμενες διαδικαστικές τροποποίησεις υπό το φως της θέσεως ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνος. Διατρέξαμε τον κατάλογο. Νομίζω αυτόν τον κατάλογο τον έχετε στους φακέλους σας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που επηρεάζεται σημαντικά ή επηρεάζεται καν από τη συνθήκη. Το βασικό που σημειώσαμε προς ενημέρωσή σας και που θα συζητήσουν αργότερα οι συντονιστές με τα ημερομηνία είναι ότι έχουμε πιο επίσημη απέτηση να έχουμε σε διαβουλεύσει με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και ζήτησα από τους συντονιστές και τη Γραμματεία να εξετάσει πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό και σε κάποιες φάσεις ίσως ζητήσουμε από εισηγητές να καλέσουν τους ομολόγους εισηγητές τους των λόγω επιτροπών να έρθουν και να μιλήσουν στη δική μας επιτροπή. Αυτό παραμένει ανοιχτό. Συμφωνείτε λοιπόν, μπορούμε να εγκρίσουμε αυτό το κείμενο omnibus και να το διαβιβάσουμε, να το κοινοποιήσουμε στη διάσκεψη των Προέδρων επισήμως. Καμία αντίρρηση. Καλώς. Θεωρείται εγκεκριμένο λοιπόν αυτός ο κατάλογος. Πάμε στην απαλλαγή του προπολογισμού 2008. Πρέπει να υιοθετηθεί για να υποβληθεί στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ο κ. Βάντερ Κάμπ ήταν ε, ο εισηγητής μας. Έχουμε τις κοιόδης κ. Γκρέπ, κ. Μπουζάρ και κ. Ρούλε. Κύριε Βάντερ Κάμπ, θέλετε να μας περιγράψετε ποιες είναι οι συστάσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και το προσωπικό για τα διάφορα σχόλιά τους και τη βοήθεια που μου έδωσαν για να ετοιμάσω την πρώτη μου τροπολογία στη δική μου ευρωπαϊκή ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε ήταν πολύ καλή η συζήτηση που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου σε μια άλλη αίθουσα. Εξετάσαμε διάφορες πτυχές του προϋπολογισμού 2008, ιδιαίτερα ε, το πρόγραμμα Solvit, πρόγραμμα Solvit και προσπαθήσαμε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του Solvit 2008 ε, στην τροπολογία που υποβάλαμε όπως τα είδατε αλλά πέραν αυτού, πέρα από αυτή την τροπολογία ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποσχεθεί σήμερα ότι θα έρθει τον επόμενο χρόνο να μας ενημερώσει για την εκτέλεση των πιστώσεων Solvit διότι αρκετοί συνάδελφοι μου το τόνισαν αυτό. Εμείς σαν Επιτροπή ΙΜΚΟ θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε να δαπανηθούν σωστά τα χρήματα του προπολογισμού για το Solvit. Αυτό είναι το σχόλιο μου αυτή τη στιγμή κύριε Πρόεδρε και βεβαίως εγώ είμαι υπέρ της ε, τροπολογίας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Συμφωνούμε πλήρως με την τροπολογία, όμως θα ήθελα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τέλος του Ιουνίου ενός τότος έτος να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση των πόρων του 2008, 2009 και 2010. Η κυρία Βερχόιβεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ. Όχι, εγώ την αντικαθιστώ. Μπορεί να μιλήσετε σε ένα λεπτάκι. Το 20% το υπόλοιπο θα πληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, λέει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας έδινα το λόγο στο τέλος, αφού ακουστούν οι άλλοι. Αλλά εφόσον απαντήσατε... Άκουσες την απάντηση Λουί ή να επαναλάβει. Άκουσα, άκουσα την απάντηση, όμως ζητούμε πλήρη έκθεση για 2008, 2009, 2010 την κατανομή των πόρων. Ας το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρο, να ακουστούν οι άλλοι σκιώδεις. Ο κ. Μποζό είναι εδώ. Δεν θα αλλάξω αυτό που είπα στην πρώτη συζήτηση. Είμαι εισηγητής για το Solvit. Λυπούμε που ξεχωριστό κονδύλι δεν είναι κρίση στον προπολογισμό. Δεν είναι νίκη για την Επιτροπή μας αυτή. Όσον αφορά την τροπολογία, υποστηρίζω πλήρως την πρώτη τροπολογία του κυρίου Βαντενκάμ, που είναι η πρώτη τροπολογία του στην ευρωπαϊκή του καριέρα και νομίζω ότι είναι και υπέρ της όλης εικόνας του Solvit που θεωρώ ότι είναι ένα αποτελεσματικό δίκτυο, αποδοτικό δίκτυο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόεδρος, η κυρία Ρούλε δεν είναι εδώ το απόγευμα. Η κυρία Γκέπχαρτ, θέλετε να μιλήσετε, ορίστε. Όχι εκ μέρου τη κυρία Ρούλε, δεν μπορεί να μιλήσω εκ μέρου τη, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφο Λουίγρεκ. Αν κατάλαβα σωστά, αυτό που απάντησε η Κομισιόν. Αυτό ουσιαστικά δεν ήταν απάντηση στην ερώτηση του Λίκρε και, και γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω το σημείο αυτό διότι είναι πολύ σημαντικό για μας τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Είχαμε τη συζήτηση για το πώς πρέπει να διατεθούν αυτοί οι πόροι. Δεν μας αρκεί να ξέρουμε ότι έχουν δαπανηθεί κατά 97% αλλά θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο να γνωρίζουμε αναλυτικά με ποιο τρόπο έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά αυτά ώστε για τον επόμενο προϋπολογισμό να μπορούμε να εξάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Right. Um, can I now... Can I now bring Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει, καταλάβατε το ερώτημα τι ζητάει δηλαδή αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή μας. Και ίσως μπορείτε να επαναλάβετε και την πρώτερη απάντησή σας. Χρησιμοποιήθηκε το κονδύλι. Χρησιμοποιήθηκε ο προπολογισμό λοιπόν για την πρόθεση του Solvit. και για την εκτύπωση εκθέσεων για την αποζημίωση των συμμετεχόντων εκπροσώπων των κρατών μελών στις ετήσιες συνεδριάσεις, στα εργαστήρια του Solvit, Solvit Workshops. Αυτά. Uh, Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να μας δώσετε ίσως πληρέστερες εξηγήσεις γραπτός με πιο αναλυτική κατανομή αν έχετε την καλοσύνη. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Uh, Επιτρέψτε να το πω στα γαλλικά για να μην υπάρχουν σφάλματα και παρεξηγήσεις. Είναι έξοχοι διερμηνείς, δεν νομίζουμε να υπάρχει πρόβλημα διερμηνίας, λέει η ομιλήτρια. Αυτό που θέλουμε το αργότερο μήνα Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει επακριβώς περί του τρόπου δαπάνης χρήσεως αυτών των χρημάτων και θα χαρούμε να δούμε τις πληροφορίες γραπτός. Αυτό είναι το απλούστερο και το καλύτερο. Αυτό που θα θέλαμε να έχουμε είναι απλώς ότι συμφωνείτε το αργότερο να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, ο ε, κύριε Κέπκατ. Ναι, απάντηση. Μπορεί να δώσει πίνακα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με λεπτομερείς αναφορές των δαπανών που έγιναν στα πλαίσια του λόγω κονδυλίου, του λόγου προπολογισμού. Καλώ λέει ο πρόεδρος, εκτός μικροφώνου. Δεν ακούμε τι λέει ο πρόεδρος δυστυχώς. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό τι ζητάμε. Προτείνω, λέει ο Πρόεδρος, να στείλω στην Επίτροπο στον Επίτροπό σας ένα σημείωμα με τις επιθυμίες της Επιτροπής μας και θα έρθω σε επαφή με τους ε, συντονιστές για να δούμε τι περιεχόμενο θέλουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα έγκριση της γνωμοδοτήσεως όσον αφορά το, την απαλλαγή του προπολογισμού. Είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Μόνο δύο ψηφοφορίε έχουμε, χρειαζόμαστε κάρτε. Τροπολογία υπαριθμών 1 του κυρίου Βάρντεν Κάμπ, παράγραφο 4 υπέρ κατά ομόφωνα ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση όλοι υπέρ κατά καλώς εγκρίνεται θα πάει στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ευχαριστούμε κύριε Κάμπ για την ομαλή διεξαγωγή αυτή της συζητήσεως με, επί της πρώτης αστροπολογίας σε αυτή την Επιτροπή ήσασταν τόσο επιτυχής που είμαι σίγουρος ότι ο συντονιστής του ΕΛΚ θα θέλει να σας δώσει πιο φιλόδοξες εκθέσεις να επεξεργαστείτε στο μέλλον. Καλώς, αυτή είναι η μόνη ψηφορία που έχουμε σήμερα. Συνάδελφοι, και καλωσορίζω στην Επιτροπή τον Ισπανό Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής ε, για τους καταναλωτές, τον κύριο Φρανσίσκο Ζαπατέρο, Φρανσίσκο Μόζα Ζαπατέρο, τον καλωσορίζω και του ζητώ να μας μιλήσει για τις φιλοδοξίες της Ισπανικής Προεδρίας όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια που είναι στον έλεγχό του και όσον αφορά τα θέματα που εξεργαζόμαστε εμείς, κυρίως δικαιώματα για τους δικαιώματα καταναλωτών, κλωστοϊφαντουργία, ονομασία στην κλωστοϊφαντουργία κλπ. Και άλλα θέματα σας ενδιαφέρουν. Οι συντονιστές συναντήθηκα με την Υπουργό σα και έχει αρκετά ενδιαφέρουσε ιδέε από ό,τι γνωρίζω, όπω όπως αποκλεισμό και επαφή συμμετοχή των καταναλωτών που σας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν και την Επιτροπή και ελπίζω να μας ενημερώσετε και ελπίζω ε, να θέλουν και συνάδελφοι συμμετάσχουν σε λόγο πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι έτσι ετοιμάσαμε το σκηνικό, οπότε σας καλώ να μας μιλήσετε και μετά θα ανοίξει ο κατάλογο ομιλητών. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι θα ήθελα να σα θέσουν κάποιε ερωτήσει. Κύριε Ζαπατέρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι αναλαμβάνει την εξάμενη Προεδρία η Ισπανία με μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να δουλέψουμε δραστήρια για όλα τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σχέδιο που είναι κοινό για όλους μας. Θέλουμε περισσότερη κοινωνική πρόοδο και οικονομική πρόοδο. Αντιλαμβανόμεθα ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία αυτή μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που τώρα ξεκινάει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Μια συνθήκη η οποία προσφέρει περισσότερη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέσα για να αντιμετωπίσει καλύτερα της προκλήσεις του μέλλοντος για ένα νέο ευρωπαϊκό κύκλο. Με αυτή τη νέα συνθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά νέες αρμοδιότητες οι οποίες θα μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο να ολοκληρώσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όλα αυτά όμως δεν θα τα πετύχουμε παρά μόνο ε, φροντίζοντας να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των πολιτών των 27 χωρών και από την άλλη μεριά την εσωτερική αγορά. Πρέπει να είμαστε σε θέση να συνδυάσουμε την εσωτερική αγορά με υπηρεσίες οι οποίες να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη μεριά οι πολίτες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να μπορούν να υποφελούνται από βασικά δικαιώματα να μην έχει σημασία σε ποια χώρα βρίσκονται, σε ποια χώρα δουλεύουν, σε ποια χώρα αποκτάνε υπηρεσίε και αγαθά. Τα δικαιώματά του πρέπει να τηρούνται πάντα. Μόνο τότε θα νιώσουν εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολλέ οι πτυχέ που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Προεδρία, δηλαδή την Ισπανική κυβέρνηση. Τα δικαιώματα όσον αφορά ε, μάλλον η όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη διακρίνεται ακριβώ επειδή έχει ένα κοινωνικό μοντέλο. Το ξέρετε, το επενθύμησε και ο πρόεδρο, Η κοινωνική πολιτική είναι πολύ βασική για την κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποτελεί ένα παράδειγμα πρόθεσης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Για να συνεχιστεί αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι ίδιοι καταναλωτές πολύ καλά τα δικαιώματά τους. Όσον αφορά λοιπόν τη σχετική οδηγία, η ΟΚΕ, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και κάποια κρατή-μέλη θέλουν μια μέγιστη εναρμόνιση. Κάτι το οποίο όμω δημιουργεί δυσκολίε όσον αφορά την εφαρμογή σε διάφορε χώρε. Ορισμένε χώρε το είπανε και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Ορισμένες λοιπόν έχουν αφιβολίες για το σε ποια θέση θα βρεθούν οι καταναλωτές εφόσον εφαρμοστεί ένα τέτοιο ε, κείμενο. Η Προεδρία μας συμφωνεί για μια εσωτερική αγορά χωρίς εμπόδια για τους καταναλωτές. Όμως πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Η οδηγία αυτή λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, όπως λέει και η συνθήκη, και να σέβεται την επικουρικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και είναι αναγκαίο να φροντίσουμε να έχουμε κάποια περιθώρια. Χρειάζεται ένα περιθώριο, να επιτρέψουμε δηλαδή στις διάφορες χώρες να αποφασίσουν μόνες τους πώς θα προχωρήσουν. Αυτός είναι ένας στόχος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ισπανία. Η θέση της Προεδρίας είναι συνένεση βέβαια, δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Πέρα από οποιαδήποτε θέση υποστηρίζει η Ισπανία, εμείς ως Προεδρία θα προτείνουμε τα μέτρα και τις συμφωνίες έτσι ώστε να επιτευχθεί συνένεση στη συνέχεια. Θέλουμε διάλογο και θέλουμε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε όλους. Είναι δικιά μας ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Να ακούσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ακούσουμε τους εργοδότες, επιχειρηματίες, τους καταναλωτές και όλοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ένα διάλογο ο οποίος θα μας οδηγήσει στη συνένεση και στην έγκριση τελικά της οδηγίας αυτής. Ίσως θα πρέπει και να δούμε ε, κάπως τι δυνατότητες υπάρχουν μικτής εναρμόνισης. Δεν λέω ότι αυτή είναι η τελική θέση, όχι. Αλλά μετά από τόσα ακούσαμε στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου, φαίνεται η μεικτή εναρμόνιση να είναι ένας εναλλακτικός δρόμος ας τον δούμε. Αντί για τη μέγιστη εναρμόνιση στα κεφάλαια, στους τίτλους εκείνους που υπάρχει συμφωνία, εντάξει, μέγιστη εναρμόνιση, αλλά να δούμε μήπως έχουμε διαφορετική εναρμόνιση στα υπόλοιπα κεφάλαια. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, λέω ότι είναι μια δυνατότητα που έχουμε μπροστά μας. Αυτή η μεικτή εναρμόνιση είναι μια θέση που στο τελευταίο Συμβούλιο ε, έχει τη συνένεση πολλών χωρών και συνάδει με την ε, αγορά. Γι' αυτό λοιπόν το εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τις υποχωρήσεις που χρειάζονται ώστε να καταλήξουμε τελικά να υιοθετήσουμε τη σχετική οδηγία. Γι' αυτό και για μας η Προεδρία δεν πρέπει να είναι εξάμεινη. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είναι μια συντονισμένη Προεδρία 18 μήνου. Έτσι μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Με το συντονισμό λοιπόν μεταξύ των διαφόρων προεδριών των εξαμήνων πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε επιτυχία. Έχουμε τώρα στην υφαντουργία, στη σχετική νομοθεσία, έχουμε μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει η συζήτηση επί Ισπανικής Προεδρίας. Όπως ξέρετε, στόχος είναι η απλοποίηση των ε, ρυθμίσεων που ισχύουν όσον αφορά τα κλειστοϊφαντουργικά προϊόντα ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να υποφεληθούν πιο εύκολα από καινοτόμα προϊόντα. Η κοινή θέση στο Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ότι έχει επιτευχθεί λίγο πολύ από τον Νοέμβριο. Μπορεί να υπάρχουν κάποια λίγα κενά, αλλά υπάρχει γενικά κοινή θέση στο Συμβούλιο. Με τη συμφωνία της Κομισιόν μάλιστα, η οποία επαφείται στον εισηγητή. Έχουμε προγραμματίσει και στις 16 Φεβρουαρίου μία επόμενη συνάντηση και μία άλλη το Μάρτιο ώστε τελικά να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών χωρών όσο γίνεται πιο γρήγορα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Τρίτος άξονας, πριν περάσουμε σε άλλα θεματάκια, είναι η δικιά μου αρμοδιότητα της ασφάλειας των προϊόντων. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τη σχετική οδηγία για την ασφάλεια προϊόντων. Δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί απαραίτητα αυτό το εξάμεινο, αλλά για μα είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί έχει άμεσε επιπτώσει στον πολίτη. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία τη κοινή γνώμη για όλα όσα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ε, μηχανισμοί ε, άμεσης αντίδρασης, το σύστημα RAPIX το καμπανάκι του συναγερμού στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα τρόφιμα, για παράδειγμα. Θέλουμε λοιπόν καλύτερο συντονισμό και με τις τελωνιακές αρχές. Να μπορούμε να βρίσκουμε τα ίχνη των προϊόντων και να χρησιμοποιείται περισσότερο τυποποίηση για να είμαστε βέβαιοι για την ασφάλεια των προϊόντων. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια διάσκεψη για την ασφάλεια των προϊόντων στη Μαγιόρκα μέσα στις επόμενες μέρες 10 και 11 Ιουνίου. θα σας προσκαλέσουμε γιατί θα ήταν καλό να υπάρχει η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί ώστε ήδη από την αρχή τη συζήτηση για την αναθεώρηση των σχετικών ρυθμίσεων να συμμετέχετε κι εσείς. Στη διάσκεψη αυτή θα μελετήσουμε εκτός άλλου και άλλου τρόπους αξιολόγησης κινδύνου για τα προϊόντα από όλες τις αρχές που ασχολούνται με την ασφάλεια των προϊόντων. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τους παραγωγούς και αυτούς που κάνουν τη διανομή των προϊόντων και να δούμε μήπως καταλήξουμε και σε τροπολογίες. Χοντρικά αυτοί είναι οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα δουλέψει η Ισπανική Προεδρία. Θέλουμε τη δικιά σας τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες. Και είναι πολύ βασικό αυτό όταν σχεδιάζουμε πολιτικές για τους πολίτες. Η γνώμη των πολιτών και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους πολίτες για την Ισπανική Προεδρία είναι κάτι ζωτική σημασία προκειμένου να γνωρίζουμε τα, ποια είναι τα προβλήματα και να εντοπίσουμε τα προβλήματα στα οποία καλούμεθα να δώσουμε λύση με αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο κλειδί στις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο λοιπόν που μου διαθέσατε. Είμαι τώρα στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Well, thank you very much indeed. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Ακούσαμε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ιδιαίτερα την ανακοίνωσή σας για την ασφάλεια των προϊόντων, στην οποία θα θέλουν να αναφερθούν οι συνάδελφοί μας. Θα ήθελα καταρχήν να καλέσουν να καλέσω τους συντονιστές μας, ε, τον κύριο Σφάπτε, τον κύριο Κέπχαρτε και τον κύριο Πουζόη. Ε, ο κύριος Πίλαν δεν είναι εδώ. Και μετά θα ανοίξουμε τη γενική συζήτηση. Ε, ο κύριος Πάρκης, ο κύριος Ροσφόρο έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Παπάκης. Ο κύριος Σφάπ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, θα ήθελα καταρχήν εκ μέρους του ΕΛΚ να σας ευχαριστήσω για την ετοιμότητά σας να εμφανιστείτε γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Ε, η Ευρώπη, ε, δεδομένη στις ε, συνθήκες της Λισαβόνας, εξαρτάται όλο και περισσότερο από το να λαμβάνονται αποφάσεις ευρωπαϊκές στο Συμβούλιο. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που είσαστε διατεθειμένους να προωθήσετε την Ευρώπη. Στην εισαγωγή σας αναφέρατε διάφορα θέματα. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο. Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ε, νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ε, το οποίο στηρίζεται. Και είμαι ευγνώμων που έχετε ένα στοχευμένο, ίσως λιγότερο φιλόδοξο ε, πρόγραμμα, αλλά ε, συγγνώμη, μια οδηγία ε, απλή, η οποία όμως να είναι πιο εύκολη στην εφαρμογή της. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω στο Συμβούλιο τι κάνετε για να πετύχετε τον στόχο αυτόν, να γίνει η οδηγία πιο ελκυστική και πιο διαφανής για τους πολίτες. και πώς μπορούμε να αποφύγουμε ε, να ε, συσσωρεύσουμε τους, ε, τις 27 νομικές τάξεις των κρατών μελών αλλά να έχουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για, που θα ωφελήσει τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις τη στιγμή που δεν είναι ακόμα σε θέση η εσωτερική αγορά να εφαρμόσει πλήρως αυτά τα στήματα θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να γίνει κάτι τέτοιο ερώτηση για την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων. Ε, πριν ε, δύο-τρία χρόνια, στα πλαίσια του πακέτου αγαθών, ε, υιοθετήσαμε μια σειρά μέτρων που από ό,τι γνωρίζω η εφαρμογή τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ήταν ήδη τότε σαφές ότι έπρεπε να λυθεί ένα θέμα που έχει να κάνει με την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων το σύστημα πληροφόρηση αναφέρθηκε ήδη στα πλαίσια του Rapid. Εμεί θέλουμε το σύστημα πληροφόρηση, αυτό να ε, λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν στην ε, ε, εισαγωγή των δεδομένων και την χρήση των πληροφοριών ώστε να μην ναυαγίσει το σχέδιο αυτό. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι σκοπεύει να κάνει η Ισπανική ε, Προεδρία για το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Κέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ Μάρκον, Ευχαριστώ πολύ κυρία Γενική Διευθυντά για την πολύ καλή εισαγωγή σας. Και εγώ χαίρομαι που ήρθατε τόσο νωρί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο έγκαιρα, για να μα δείξετε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα που έχουμε τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, την ε, οποία τονίσατε ιδιαίτερα η συνθήκη της Λισαβόνας ε, σημαίνει και ε, υψηλό επίπεδο ε, προστασίας των καταναλωτών σε συνδυασμό με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και θέλουμε προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η συζήτηση έτσι φτάνει στο θέμα της προστασίας των καταναλωτών, ε, την εναρμόνιση, τι βαθμό εναρμόνισης μπορούμε να έχουμε και σε τι επίπεδο πρέπει ή μπορεί να πραγματοποιηθεί η εναρμόνιση αυτή. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουμε να απαντήσουμε εδώ. Όταν βλέπουμε ότι στην συνθήκη της Λισαβόνας ε, δίνεται η υψηλότερη θέση στα ε, δικαιώματα του καταναλωτή, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε δρόμο ε, που να έχει ως αποτέλεσμα ε, λιγότερα δικαιώματα για τους πολίτες από ό,τι έχουν αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή όπως την έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο ψήφισμα της κυρίας Πατρί ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε ότι ε, θέλουμε μεικτή ε, προσέγγιση στην εναρμόνιση όπου είναι δυνατόν. Ε, Ευχαρίστω να έχουμε πλήρη εναρμόνιση. Αυτό αφαίρεται και στους ορισμούς, αλλά σε διάφορους τομείς το δίκαιο των κρατών μελών ε, έχει εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό μπορεί σε κάποιες χώρες ε, να έχουμε μείωση του επίπεδου προστασίας των ε, δικαιωμάτων. Και κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το δεχτούμε, διότι αυτό θα σημάνει τελικά ότι οι πολίτες θέλουν ακόμα λιγότερη Ευρώπη από ότι σήμερα. Ε, θα είναι ακόμη πιο σκεπτικιστική απέναντι στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα ήθελα να επενέσω τη συζήτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή και τον διάλογο που μας προτείνεται. Δεύτερο τομέα που θέλω να αναφέρω, ε, δεύτερο τομέα που θέλω να αναφέρω είναι τα υφάσματα. Ε, μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Σβάπ. Πράγματι, θέλουμε απλοποίηση του δικαίου όσον αφορά την έγκριση νέων προϊόντων. Ωστόσο και εδώ θα πρέπει η προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια των καταναλωτών ε, να έχουν προτεραιότητα. Και πρέπει να πω ότι η συζήτηση αυτή εμένα προκαλεί ένα περίεργο συνέστημα, διότι θα πρέπει να εμποδίσουμε ή όχι, διότι η συζήτηση αυτή έχει το χρώμα αν θα πρέπει ή όχι να εμποδίσουμε τι τις επιχειρήσεις να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όταν οι επιχειρήσεις αποφάσισουν να λανσάρουν στην αγορά νέα προϊόντα, να ε, είναι ασφαλή τα προϊόντα αυτά. Και η δική μου πολιτική ομάδα δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση της ασφάλειας ε, των πολιτών και αυτό είναι χρέος των ε, επιχειρήσεων να το φροντίσουν αυτό όταν ε, διαθέτουν στην αγορά νέα προϊόντα, διότι άλλωστε βγάζουν χρήματα από αυτό. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο. Τελευταία παρατήρηση και συγγνώμη που μακρηγορώ εφαρμογή της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και μεταξύ των συντονιστών έχουμε λάβει σχετική απόφαση και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Με τα Εθνικά Κοινοβούλια θέλουμε να συζητήσουμε και την εφαρμογή ε, της οδηγίας αυτής και ε, τα ενδιαφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή τους επόμενους μήνες και θα είμαι ευγνώμων εάν ε, η Προεδρία του Συμβουλίου ε, παρακολουθήσει στενά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Διευθυντά, βλέπετε ότι καλύπτουμε πολλά διάφορα θέματα. Ο κύριος Πουζόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμάνικα. Κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Έχουμε υψηλές προσδοκίες από την Ισπανική Προεδρία η οποία ξεκινάει σε μια χρονική στιγμή που η αρχιτεκτονική της Ευρώπης έχει νέα θεμέλια, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μιλήσατε για την προστασία των καταναλωτών και παρακολούθησα στενά αυτά που είπατε. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2010. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα αφήσω το λόγο στον συνάδελφό μου τον κύριο Ροσφόρ που είναι σκιώδης εισηγητής της ομάδας των φιλελευθέρων. Αλλά θα ήθελα να πω λίγα λόγια. Προέρχομαι από νέο κράτος μέλος και ξέρω ότι ο κόσμος έχει διαφορετικές εμπειρίες με την ομοθεσία στον τομέα αυτών. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες που προσπαθούν, τους οποίους προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και που έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα θέματα σε διάφορα κρατημέλη, αλλά επηρεάζονται και οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να προσαρμοστούν στις διάφορες εμπειρίες και τις διάφορες νομικές τάξεις που απαντούν όσον αφορά την προστασία των ε, καταναλωτών στα διάφορα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο να γίνει ρύθμιση υψηλού επίπεδου για κάθε λεπτομέρεια του τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Πιστεύουμε ότι η μεικτή εναρμόνιση αποτελεί σωστή λύση. Θα σας παρακαλούσα όμως να μου πείτε εάν η Ισπανική Προεδρία στηρίζει την αρχή της ε, μικτής εναρμόνισης να μου πείτε εάν στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, εάν έχετε προτάσεις τροποποίησης και αν ναι, ποιες είναι αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουζόη. Να δώσω το λόγο στους βουλευτές. Έχω τον κύριο Πουπάκη και τον κύριο Ροσφόρ. Είναι ανοιχτός ο κατάλογος των νεομιλητών εάν θέλει κάποιος άλλος να παρέμβει. Ο κύριος Πουπάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και το Γενικό Διευθυντή για την διάθεσή του να ενημερώσει και μάλιστα άμεσα Διαβάζοντας προσεκτικά το συνολικό πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας, θα ήθελα να σας συγχαρώ, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιους τομεί που έχει ανάγκη η κοινωνία, όπως η οικονομία, η τόνωση τη ανάπτυξη και της απασχόλησης. Ωστόσο φοβάμαι ότι η κοινωνική ατζέντα λόγω της οικονομικής κρίσης, ειδικά αυτή τη στιγμή, ίσως υστερεί όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Και να συγκεκριμενοποιήσω. Εν μέσω αυτή λοιπόν της κρίσης, όταν το 17% των ευρωπαίων καταναλωτών ζουν κάτω από τα όρια τη φτώχεια, εκατομμύρια καταναλωτέ προκειμένου να αντεπεξέλθουν στι δύσκολε οικονομικέ συνθήκε που αντιμετωπίζουν, καταφεύγουν δυστυχώ, μη έχοντα άλλη λύση, στο δανεισμό και στην υπερχρέωση των πιστοτικών καρτών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχουν και ποιε προτεραιότητε τη Ισπανική Προεδρία για τον υπερχρεωμένο καταναλωτή, που πολλέ φορέ γίνεται έρμεο των χαρακτηριστικών όρων των τραπεζών και ειδικότερα αν υπάρχει πρόληψη για την πρόθεση ενός σχεδίου δράσης και ενεργειών που να έχει συγκεκριμένους δύο στόχους. Πρώτον, την προστασία των κανοντών από αδιαφανείς και κερδοσκοπικές πρακτικές τραπεζών, καθώς και αμφιλογόμενα τραπεζικά προϊόντα που δυσχεραίνουν τις συνθήκες ή την προσπάθεια αποπληρωμής. Και δεύτερον, τη διασφάλωση ενός σταθερότερου και δικαιότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος με ενιαίους όρους και προϋποθέσεις που να διασφαλίζει ίση πρόσβαση και προστασία για τους δανειολήπτες Ευρωπαίους πολίτες καταναλωτές. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε ο κύριος Ροσφόρ τώρα. Και μετά κύριε Ράπτη. Ο κύριος Ροσφόρ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο γρήγορα στην αρχή της Προεδρίας σας εδώ. Βρήκα Πολύ ξεκάθαρα τα λόγια σας και χαίρομαι όταν κάποιος είναι σε θέση να μεταφέρει τις ιδέες του τόσο καθαρά. Αυτή η περίφημη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Εγώ βλέπετε είμαι καινούριο εδώ, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι ένα θέμα για το οποίο όλοι συζητάνε εδώ και πολύ καιρό. Και δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση το ότι ήσασταν έτσι ξεκάθαρος και για την επικουρικότητα και για την εναρμόνιση. Στην προηγούμενη ζωή μου βλέπετε και όταν η Γαλλία είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θυμάμαι τις εργασίες αυτές για το εμπόριο, ότι στην Ισπανία υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο ρύθμισης του εμπορίου που αφορούσε ολόκληρη τη χώρα σας και που πρόσφερε στις περιφέρειες, στις αυτόνομες περιφέρειες δηλαδή τις Ισπανίες, ελευθερίες που δεν έρχονται σε αντίθεση με την ε, λογική του γενικού δυναμισμού που υπάρχει στη χώρα σας. Τώρα να μιλάμε για μεικτή, για στοχοθετημένη ή για ανώτατη εναρμόνιση, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Και για την μεικτή εναρμόνιση να ξέρετε ότι μου αρέσει γιατί η ανώτατη εναρμόνιση δυσκολεύει τον καταναλωτή. Έχει την αίσθηση ότι θα αποκτήσει την πλήρη προστασία αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό, γιατί η εναρμόνιση έχει να κάνει μεταξύ των χωρών. Δεν έχει να κάνει με το ανώτατο επίπεδο προστασία του καταναλωτή. Εκεί λοιπόν υπάρχει παρεξήγηση. Να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί για να φτάσουμε σε κάτι που δεν θα είναι αντιφατικό, που όντω θα βοηθάει τον καταναλωτή. Όπως είπε και η κυρία Γκέπαρτ, οι ορισμοί και εδώ και αλλού πρέπει να είναι ξεκάθαροι γιατί μπορούμε ίσως να μιλάμε για χαμηλή ε, εναρμόνιση, δηλαδή μεταξύ λίγων χωρών, αλλά ανώτατη όσον αφορά το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Πάντως, στην ιδανική περίπτωση, εγώ θα ήθελα να έχουμε ένα γενικό πλαίσιο για να προστατεύουμε τον Ευρωπαίο καταναλωτή και συγχρόνως τη δυνατότητα να είμαστε ελαστικοί. Δηλαδή να αφήνουμε χώρο στην κάθε χώρα να μπορεί να εφαρμόζει και εκτιμένα δικαιώματα. Είναι δύσκολο βέβαια να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη σε μια οδηγία. Ιδίω μάλιστα όταν πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι εξελίξει, του νέου τρόπου που έχει ο καταναλωτή για να καταναλώνει. Σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια οι καταναλωτέ θα καταναλώνουν πολύ περισσότερο μέσω διαδικτύου, θα κάνουν πολύ περισσότερε αγορές online. Όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία. Και μάλιστα σήμερα το πρωί διάβαζα σε μια καθημερινή εφημερίδα κάτι για την κατανάλωση το 2009 πέρυσι. Στις περισσότερες χώρες μας όσον αφορά τα προϊόντα υψηλή τεχνολογίας, οι καταναλωτές καταναλώνουν λίγο πολύ τα ίδια για τηλεοράσει ε, υψηλή πιστότητα είτε για Blu-ray για να βλέπει κανεί ε, ταινίες με καλύτερο, καλύτερης συγκλίνει η κατάσταση στις χώρες μας. Ενώ όταν πρόκειται για τα τρόφιμα, όταν πρόκειται για τα ρούχα και πολλούς άλλους τομείς, υπάρχουν ιδιαιτερότητες στις χώρες μας και άρα διαφορές που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές και όχι τόσο με την πρακτική. Όλα αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι για τις ε, προτάσεις σας. Πώς θα συμπεριλάβετε την ανησυχία μας αυτή, δηλαδή ένα κείμενο το οποίο να είναι καλό αλλά και έτοιμο να προσαρμοστεί στις εξελίξεις, στις αλλαγές, στις καινοτομίες. Τα είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο, μίλησε για την ε, οικονομική κρίση, όντως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό και όλες αυτές οι νέες πρακτικές κατανάλωσης. Πώς θα φροντίσετε η οδηγία μας να προσαρμόζεται στις εξελίξεις κάθε τόσο. Η κύριε Ράπτη. Και ακόμα αν κάποιο άλλο θέλει το λόγο να μου το πείτε. Έχουμε λίγο χρόνο. Παρακαλώ κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. τα περισσότερα από αυτά που είχα στο μυαλό μου να πω τα είπε η Εύελιν Γκέπχαρτ. συμπληρώθηκαν πάρα πολύ ωραία και από τον κύριο Πουπάκη και από τον κύριο Ροσφόρ. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξή. Η Ισπανική κυβέρνηση και άρα η Ισπανική Προεδρία αυτή τη στιγμή είναι από τις λίγες δυστυχώς σοσιαλιστικές που υπάρχουν στο πλαίσιο της Ευρώπης. Αυτό εμένα που προέρχομαι από σοσιαλιστικό κόμμα με κάνει να ελπίζω περισσότερο. Και με κάνει να ελπίζω περισσότερο ότι θα μπορέσει να φτάσει σε ένα κείμενο οδηγίας που να είναι προς όφελος των καταναλωτών ίσως σε έναν περισσότερο μεγάλο βαθμό από ό,τι έχουμε στο μυαλό μας. Ε, επειδή συνήθως όταν έρχονται εδώ είτε υπουργοί είτε γραμματείς από τις χώρες που έχουν την προεδρία ακούμε πάρα πολύ καλές προθέσεις, ακούμε διαπιστώσεις, ακούμε αριθμούς αλλά συνήθως μένουμε ε, ανικανοποίητοι ως προς το αποτέλεσμα ε, θα παρακαλούσα ακριβώς επειδή ελπίζω πάρα πολύ στη σοσιαλιστική ισπανική προεδρία δεν θα ήθελα να μου πείτε πολλούς στόχους. Θα ήθελα να μου πείτε έναν μόνο στόχο, έναν μόνο, κανέναν άλλο, που έχετε στο μυαλό σας ότι θα θέλετε, θα θέλετε να έχετε επιτύχει στο τέλος της Προεδρίας. Έναν μόνο. Θα είμαι ευχαριστημένη και βέβαια στο μυαλό σας πάντα τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ωραία, ελπίζω να σας ικανοποιήσουμε σήμερα το απόγευμα, κύριε Ράπτη. Μια που έχουμε λίγο χρόνο, ίσως και εγώ mm-hmm. να σχολιάσω κάποια πράγματα εκ μέρους της ομάδας μου των συντηρητικών. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξέρω για τις διεθνείς προοπτικές της δουλειάς της Προεδρίας. το όραμά σα για την ανάγκη προετοιμασία για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των προϊόντων είναι πολύ καλό. Ουσιαστικά κάνετε την προπαρασκευαστική εργασία για τη διάσκεψη του Ιουνίου και ελπίζω ότι αρκετά μέλη αυτή τη Επιτροπή να μπορέσουν να παραστούν, γιατί νομίζω έτσι θέλουμε να εργαζόμαστε όπως τα παρατηρήσατε. Θέλουμε να προετοιμαζόμαστε και να συλλέγουμε πληροφορίες όταν προετοιμάζουμε ένα θέμα. Λοιπόν, υπάρχει και μια ισχυρότατη διεθνής διάσταση όσον αφορά την ασφάλεια ε, των προϊόντων και σε παγκόσμιο επίπεδο των προϊόντων που εισάγονται στην ενιαία αγορά και αυτή η Επιτροπή ε, το 2008 ασχολήθηκε πολύ με την Κίνα. Πήγαμε σε αποστολή εκεί και εξετάσαμε κάποια τα θέματα και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. επικεφαλής της η κυρία Τάνενμπαουμ, που είναι Αμερικανίδα επικεφαλή τη Επιτροπή για την Ασφάλεια Προϊόντων για του Καταναλωτέ, ζήτησε να έχουμε μια τηλεδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω οι συντονιστέ να μπορούν να έρθουν. Δυστυχώ δεν μπορεί να έρθει όλη η Επιτροπή, γιατί έχουμε μικρή αίθουσα διαθέσιμη για βίντεο διασκέψει. Λοιπόν, εσεί διεθνώ, τι στόχο έχετε, πώ βλέπετε να προχωράει, και ίσω για τη ίσω να έχετε υπόψη να προσκαλέσετε κάποιον από την Επιτροπή Ασφαλείας Προϊόντων των ΗΠΑ ή από την Κίνα να έρθουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα, διότι έχει ε, διεθνή διάσταση και παγκόσμια διάσταση αυτό το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ήθελα να σας δείξω αφορά παλιές εργασίες αυτής της Επιτροπής μας, διότι μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε και άλλες εργασίες με τις οποίες έχουμε διασυνδεθεί και να δούμε πώς υλοποιούνται όλα αυτοί οι στόχοι και ενδιαφέρεται πολύ και το Συμβούλιο και στο πρόγραμμα του Συμβουλίου θα θέσετε διάφορα θέματα που αφορούν την εφαρμογή σε εθνικό δίκαιο διαφόρων βασικών οδηγιών. Κάτι που πιθανά εμπίπτει στις ευθύνες σας στο Συμβούλιο είναι η οδηγία για την ε, καταναλωτική πίστη, για τις πιστώσεις για τους καταναλωτές. Ο κύριος Ρόσφορ απέθυνε μια ε, ένθερμη έκκληση να δούμε αν πρέπει να είναι μεικτή ή εστιασμένη εναρμόνιση στα δικαιώματα των καταναλωτών ή καμία εναρμόνιση ή να εναρμονιστούν κάποιοι τομεί. Η οδηγία λοιπόν για αυτή την καταναλωτική πίστη είναι ακριβώ ένα θέμα ε, στοχευμένη εναρμόνισης και εμεί αντίθετα από αυτά που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν Επιτροπή αποφασίσαμε τα δικά μα. Και αντικατοπτίζεται αντικατοπτρίζεται αυτό και στην οδηγία για τα δικαιώματα καταναλωτών υπήρχαν κάποια στοιχεία καταναλωτικής πίστης και οι παραδόσεις προϊόντων στους καταναλωτές πρέπει να εναρμονιστούν στα κράτη-μέλη και κυρίως όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν συνάδελφοι το απόγευμα περί δυνατότητας ε, αποπληρωμής δοθέντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το θέμα της χρέωσης των χρεών μαζί με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στη διεύθυνση εσωτερικής αγοράς. Κατά πόσο δίνεται συνέχεια σε αυτό. Και όταν μιλούσα σε διασκέψεις και ακροάσεις όσον αφορά τα χρέη αυτά, κάποια στοιχεία που ήταν στην οδηγία για καταναλωτική πίστη μπορούσαν να ενταχθούν σε θέματα ε, ιδιοκτησίας ε, εσωτερικής κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποια από αυτά εμπίπτουν στις δικές σας αρμοδιότητες. Αυτή είναι η δική μου συνεισφορά. Η κυρία Γκέπχαρτ θέλει να δευτερολογήσει με τα χαράς και μετά θα σας δώσω το λόγο σε εσά κύριε Γενική Γραμματεύκο. Πρώτα η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρθηκε η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και θυμήθηκα κάτι πολύ σημαντικό η οδηγία αυτή ισχύει μόνο από ένα συγκεκριμένο ποσό και πάνω και δεν το θυμάμαι το ποσό αυτό. Ο συνάδελφος Μητρορέπο πέσε την προσοχή μας σε ένα πρόβλημα. Ότι όλο και πιο συχνά χορηγούνται μικρές πιστώσεις, μικροπιστώσεις, ε, όχι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά και με SMS. Και οι πελάτες ε, συχνά είναι πολύ νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται ότι μπορεί να υπερχρεωθούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και βλέπω ότι ο κύριος Μπαρνιέ, ο μελλοντικό επίτροπος για την εσωτερική αγορά, είναι παρόν. Ε, ίσως να μπορεί να ακούσει και αυτός τι έχω να πω. Είναι επίγον το θέμα. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση θα πρέπει να βρούμε μια απάντηση στο θέμα αυτό, διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε νέοι άνθρωποι να ε, μπαίνουν σε πολλά χρέη και ε, την υπόλοιπη ζωή τους ε, να πληρώνουν ένα λάθος που έκαναν από άγνοια. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό. Δεν ξέρω με ποια μορφή, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έθιξε και η σουηδική κυβέρνηση απέναντί μας. 200 ευρώ είναι το κατόφλι. Ωραία. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους, ε, κύριε Γενική ε, Γραμματέα, κύριε Γενική Διευθυντά. Θα παρακαλούσαν να πάρετε το λόγο και να απαντήσετε σε, στις ερωτήσεις αυτές και να κάνετε και άλλες ενδεχομένως παρατηρήσεις ε, για σήμερα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνεκτικά και σύντομα και συγκεκριμένα. Πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν που μερικές ήταν ε, πολύ κοντά μεταξύ τους. Οπότε θα τις συγκεντρώσω αυτές. Για την οδηγία. Ο κύριος Σουάπ για την οδηγία όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών ρωτάει τι θα κάνουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού και όχι προσθέτοντα το τι ισχύει στι διάφορε χώρε. Ο στόχο μα πρέπει να είναι διτό. Από τη μια μεριά η εσωτερική αγορά, να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη εναρμόνιση μέσα στην εσωτερική αγορά για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλο και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσεί με αυτό που είναι να μην περιοριστούμε σε δικαιώματα που ήδη είναι κεκτημένα. Θα ήταν πολύ περίπλοκο να εξηγήσουμε στον καταναλωτή και να του πούμε ότι μέχρι τώρα μπορούσατε να επιστρέφετε ένα προϊόν που έχετε αγοράσει χωρίς κανένα όριο. Τώρα με την οδηγία η οποία ισχύει για να βελτιωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, ε, τώρα πια δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Ε, καταλαβαίνετε, δεν το καταλαβαίνει αυτό ο καταναλωτή. Όταν έχει κάποιε εγγυήσει διαβίου για ένα προϊόν ο καταναλωτή, και τώρα το πούμε όχι, ισχύει μόνο για δύο χρόνια και τον τρίτο χρόνο δεν γίνεται, γιατί η Ευρώπη έτσι αποφάσισε, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολο. Το... Η Ευρώπη που φτιάχνουμε δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση στους καταναλωτές ότι περιορίζουμε τα δικαιώματά τους. Το αντίθετο. Είναι δικιά μας ευθύνη λοιπόν της Προεδρίας αλλά και της Κομισιόν να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και να δείξουμε ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές. Και όλοι σας αυτό ζητήσατε. Ζητήσατε μία μεικτή εναρμόνιση. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να πάρω θέση ως Προεδρία αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι ως Προεδρία οφείλουμε να βοηθήσουμε να επιτευχθεί συμφωνία. Αν τώρα ε, το Συμβούλιο συνεχίσει όπως και μέχρι τώρα έκανε, τότε εκεί θα καταλήξουμε. Στην μεικτή εναρμόνιση δεν βλέπω άλλη δυνατότητα, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων. Εδώ υπάρχουν νέοι στόχοι στην αναθεώρηση αυτή και ένας είναι εναρμόνιση με τον κανονισμό για να μην υπάρχουν ανομαλίες, να απλοποιήσουμε τη διαδικασία τυποποίησης ώστε να είναι πιο απλή, να ενισχύσουμε την κλεισιμότητα των προϊόντων συμπεριλαμβάνοντας αυτό που λέει και ο κανονισμός, να αναθεωρήσουμε τη, τα προσωρινά μέτρα, να βελτιώσουμε το διοικητικό συντονισμό εποπτείας, να ενσωματίσουμε την οδηγία για την εξαπάτηση, να μελετήσουμε την παρακολούθηση online διαφόρων προϊόντων, να ξαναδούμε την ασφάλεια των προϊόντων και να εισαγάγουμε και μηχανισμούς για τη συλλογή στοιχείων όσον αφορά τον έλεγχο της αγοράς σε σχέση με το RAPEX. Τρεις δρόμοι δηλαδή. Απλοποίηση του όσου υπάρχουν, ε, απλοποίηση και να δούμε πώς μπορεί να γίνει παρακολούθηση online. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τις νέες τεχνολογίες για να έχουμε τα ίχνη των προϊόντων. Πάνω σε όλα αυτά τα στοιχεία θα δουλέψουμε μαζί, θα συνεργαστούμε. Στη Μαγιόρκα πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά και να προχωρήσουμε συντονισμένα με τη βιομηχανία, με τους καταναλωτές και με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η κυρία Γέπαρτ με ρώτησε για την προστασία των καταναλωτών πώ θα γίνει να μην περιοριστούν τα δικαιώματά του. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορούμε, όπω είπα και πριν, να φτιάξουμε την Ευρώπη περιορίζοντα τα δικαιώματα η αναρμόνιση πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Στο κάτω-κάτω μπορεί να μην μπορέσουμε με μία οδηγία να πετύχουμε την αναρμόνιση που θέλουμε, αλλά δεν πρέπει κανένας πολίτης να νιώθει ότι πάμε πίσω αντί να πηγαίνουμε μπροστά. Από ό,τι έχουμε δει στα πρόσφατα συμβούλια, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε συγχρόνως ότι χρειάζεται τυποποίηση της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να ζυγίζουμε αυτά τα δύο. Μικτή εναρμόνιση είναι ο καλύτερος δρόμος, μου φαίνεται. Για την υφαντουργιά. Είπαμε ότι έχουμε συμφωνία λίγο πολύ πάνω στο κείμενο. Θα βελτιωθεί η ευελιξία του πλαισίου προστατεύοντας τους καταναλωτές. Ο κανονισμός ο ίδιος μας προσφέρει επιχειρήματα για να βάλουμε μπρο νομοθεσία και για άλλα θεμελιώδη ζητήματα. Τα αλλεργιογόνα, η μελέτη των αλλεργιογόνων για παράδειγμα, απαιτεί μια πολύ καλή μελέτη, η οποία πρέπει να πάρει το χρόνο που χρειάζεται για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Όλοι θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση ξεκινώντας από την μελέτη για τα λεριογόνα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την προστασία του καταναλωτή. Αναμφίβολα, ό,τι μελετάμε για τις νέες ίνες χρειάζεται να καταλήξει σε μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή. Αυτό είναι το νόημα. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για την πίστοση των καταναλωτών. Είναι πράγματα τα οποία προχωράνε σε διάφορες χώρες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανησυχία. Ίσως θα ήταν καλό η Κομισιό να μας πει περισσότερα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, τις υπερχρέωσεις κλπ. Καταλαβαίνω την ανησυχία που υπάρχει. Και είμαι σίγουρος ότι η Κομισιόν θα μας βοηθήσει για να προχωρήσουμε ο κύριος Μπουσόη. Για την εναρμόνιση τη μεικτή. Δεν θέλω εδώ να τοποθετηθώ, αλλά έτσι όπως φάνηκε από τις τελευταίες συνεδριάσεις στο Συμβούλιο, είναι πιο εύκολο να καταλήξουμε για ορισμένους σε πλήρη εναρμόνιση, άλλοι θέλουν άλλου είδους εναρμόνιση μη περιοριστική για τις χώρες. Κατά πάσα πιθανότητα, τρία κεφάλαια βλέπουμε να έχουν προσέγγιση των θέσεων για πλήρη αναρμόνιση και τα κεφάλαια που έχουν να κάνουν με την αναρμόνιση δικαιωμάτων ή δικαικτημένων από τους καταναλωτές, ή τους καταναλωτές είναι κάτι πιο περίπλοκο και πιο δύσκολο να βελτιωθούν τα δικαιώματα στις χώρες μέλη αλλά πρέπει να το μελετήσουμε περισσότερο. Ως Προεδρία θα προσπαθήσουμε να σφιγμομετρήσουμε κάπως το Συμβούλιο για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Για τον κύριο Πουπάκη. Συμφωνώ απόλυτα με πολλά από αυτά που είπατε. Και επιπλέον Υπάρχει και η κοινωνική πολιτική και η κατανάλωση και τα δύο είναι δικά μου θέματα. Είμαι πεπισμένο ότι οι περίοδοι κρίσης δεν πρέπει να χρησιμεύουν για περιορισμό των δικαιωμάτων των πολιτών και κυρίως των πολιτών ω καταναλωτέ. Κάθε άλλο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα σε ποια στιγμή βρισκόμαστε σήμερα για να προωθήσουμε τα δικαιώματά τους. Εδώ βέβαια η συζήτηση είναι ευρύτερη τι διαφεροποίηση μπορούμε να προσφέρουμε. Αυτό πρέπει να έχει να κάνει με την ποιότητα, όχι με τον περιορισμό των δικαιωμάτων. Και σίγουρα πρέπει να δείξουμε ευαισθητοποίηση σε όλα αυτά που είπατε. Είναι και το έτος καταπολέμησης της ένδυας και του κοινωνικού αποκλείσμου. Δεν είναι τυχαίο. Έχουμε δεκατομμύρια ανθρώπους που κινδυνεύουν με ένδυα και πρέπει να τους διασφαλίσουμε κάποιο επίπεδο έτσι ώστε να τους δώσουμε τη σιγουριά ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή η κατάσταση. Η στρατηγική 2020 είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της κοινωνικής ε, περιθωριοποίησης, του κοινωνικού αποκλεισμού. Βέβαια, η στρατηγική αυτή πρέπει να συμπεριλάβει και θέματα καταναλωτών και δικαιωμάτων καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα το τραπεζικό σύστημα, από πλευρά της κατανάλωση. μιλάμε για την μεταρρύθμιση. Από πλευρά τη κυβέρνησή μου, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο μπαίνει στη συζήτηση, το άκουσα χτε αυτό για τον κύριο Ροσφόρ. Για την επικουρικότητα μιλήσατε. Όντως, υπάρχει πλήρης αποκέντρωση στην Ισπανία. Αυτό είναι αλήθεια. Εντόπισα σημαντικά πράγματα σε αυτά που μας είπατε. Πρώτα απ' όλα το θέμα της ελαστικότητας, έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις εξελίξεις στην πρόοδο των νέων τεχνολογιών για να μην μένουμε πίσω. Αναφίβολα αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει εγκάρσια να δούμε για την προστασία των καταναλωτών. Πριν αναφερθήκαμε στην ασφάλεια των προϊόντων και την πώληση μέσω ίντερνετ. Πρέπει να μπορούμε να βρούμε τα ίχνη των προϊόντων για να είμαστε σίγουροι για την ασφαλειά τους. Πιστεύω ότι η ελαστικότητα πρέπει να υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις και να απορρέει από την ε, μεικτή εναρμόνιση. Συγγνώμη που αναφέρομαι στην ισπανική περίπτωση, αν και εδώ εκπροσωπώ την Προεδρία, αλλά θέλω να σας απαντήσω. Εμείς Μπορεί να έχουμε μια συγκεκριμένη εναρμόνιση που να επιτρέπει μια αυτόνομη περιφέρεια να μπορεί να πάει όμως πιο πέρα, να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη προστασία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτό πρέπει να το συνδυάζουμε με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη χώρα, στην αυτόνομη περιφέρεια και την ευρωπαϊκή ρύθμιση. Κοιτάξτε, ως ε, Προεδρία δεν μπορώ να αναφερθώ στην Ισπανική κυβέρνηση, τη σοσιαλιστική, αλλά για το αποτελέσμα, για το στόχο που με ρωτήσατε κύριε Ράπτη. Είναι περίπλοκο. Αλλά καταλαβαίνω σε έξι μήνες θα είναι πολύ εύκολο να πείτε αν τα κατάφερε ή δεν τα κατάφερα ως Προεδρία. Τι να πω. Αν θέλω να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη, θα έλεγα να έχουμε ένα κείμενο όσον αφορά τον κανονισμό για την υφαντουργία. Να, Και μετά τι θα μου πείτε, περάσατε ή δεν περάσατε τις εξετάσεις. Να. Αλλά υπάρχει και κάτι πιο θεμελιώδες. Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών να είναι τέτοια που να διασφαλίζει ότι κανενός Ευρωπαίου πολίτη καταναλωτή τα δικαιώματα δεν θα μειωθούν. Είναι μια θέληση, μια βούληση που έχουν και όλες οι χώρες και όλα τα θεσμικά όργανα. Η βούληση υπάρχει. Αλλά από αυτά που είδα στα τελευταία συμβούλια, η βούληση υπάρχει. Κανένας καταναλωτής να μην ε, δει τα δικαιώματά του να περιορίζονται μέσα από τα νέα κείμενα στο οποίο θα καταλήξουμε. Η δικιά μας η δουλειά ως Ισπανική Προεδρία είναι να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε με τις δύο προεδρίες ώστε τα αποτελέσματα Μπορεί να μην είναι στην Ισπανική Προεδρία, να είναι στη Βέλγια και στην Ουγγρική, αλλά να είναι όσο γίνεται πιο θετικά. Η δικιά μας ευθύνη είναι να βλέπουμε τα πράγματα με κάποια προοπτική. Ελπίζω να προχωρήσει η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το στοιχείο κλειδί, γύρω από το οποίο θα στραφούν πολλές αποφάσεις για τα μελλοντικά δικαιώματα των καταναλωτών, θα είναι αυτή. Κύριε Χάρμπορ, για το πώς θα βρεθείτε στη Μαγιόρκα, το έπιασα το μήνυμα. Θα σας στείλουμε προσκλήσεις για να μπορέσετε να έρθετε. Στο, σας το γιώμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ήδη από την αρχή της συζήτησης και τώρα είναι η αρχή της συζήτησης να εκπροσωπούνται όλα τα θεσμικά όργανα. Στην προηγούμενη συνάντηση όταν είχαμε κάποια άτυπη επαφή μαζί σας, υπουργό και εγώ, είπαμε ότι πρέπει να έχουμε αυτή τη συνεργασία για να καταλήξουμε πιο εύκολα σε αποτελέσματα. Είναι θέμα λογικής. Με τα εθνικά κοινοβούλια το κάνουμε. Είναι το σύνηθες, ήθιστε. Είναι πρακτική που ακολουθούμε. Η συνάντηση στη Μαγιόρκα λοιπόν, πέρα από μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία που θα έχετε για να αποφεληθείτε από τις βαλερίδες νήσους μέσα στον Ιούνιο που είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου γι' αυτό, είναι επιπλέον μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να δουλέψουμε και να ενισχύσουμε και τα προϊόντα, την προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματά τους, αλλά και ε, την ε, ποιότητα των προϊόντων και την ασφάλεια των προϊόντων. Και οι Κινέζοι θα είναι και άλλες χώρες θα καλέσουμε προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα της ε, χνηλασίας των προϊόντων και προκειμένου επίσης να συντονίσουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να εντοπίζουμε κινδύνους. Θέλουμε να έχουμε ένα ευρύ δίκτυο. Να μην βασιζόμαστε μόνο στο σύστημα συναγερμού το ευρωπαϊκό. Θέλουμε να έχουμε συντονισμό ευρύτερο. Και η Κομισιόν και διμερός προσπαθούμε να το πετύχουμε. Είναι πολύ βασικό για μας για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των προϊόντων η βούληση υπάρχει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε και οι ΗΠΑ και η Κίνα και άλλες πλευρές να συμμετέχουν στην ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η στρατηγική μας πρέπει να είναι συντονισμένη και σφαιρική. Για τις πιστώσεις απάντησα για τη σχετική οδηγία της καταναλωτικής πίστης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εμπεριστατωμένη αυτή παρουσίαση. Μα στείλατε μηνύματα για τα δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι σημαντικό για τον κύριο Σβάμπ αυτό, σαν μήνυμα, που περιμένουμε επίση να ετοιμάσει την έκθεσή του κατά την Προεδρία σα. Είναι ένα έγγραφο που περιμένουμε ανυπόμονα και θα το συζητήσουμε εκτενώς και λεπτομερώς. Καλωσορίζουμε και τη δέσμευσή σα για διάφορα θέματα. Και όταν μιλήσω με την κυρία Τάνενμπαμ την επόμενη εβδομάδα θα την ενθαρρύνω να έρθει η ίδια στην διάσκεψη για την ασφάλεια των προϊόντων ή να εκπροσωπηθούν οι ΙΠΑ τουλάχιστον. Θα σα το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ικανοποίησατε. Είναι χαρούμενη η κυρία Ράπτη. Τη βλέπω να χαμογελάει. Είναι ευχαριστημένη με τι δεσμεύσει που αναλάβατε. Σας ευχόμεθα ότι καλείτε την Προεδρία σας. Θα στείλουμε αντιπροσωπεία στην Ισπανία σε τρεις εβδομάδες. Δυστυχώς έχω οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν θα έρθω, αλλά διάφοροι συνάδελφοι θα έρθουν. Οπότε ίσως έχουμε την δυνατότητα στη Μαδρίτη να συναντήσουμε και εσά και το προσωπικό σας. Θα πάμε και στο Αλικάντε, οπότε αυξάνουμε τις προσπάθειές μας. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ για την δουλειά σας και σίγουρα και οι συνάδελφοί μου όπως και εγώ θα σας ευχηθούμε καλή τύχη με την Προεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Yes, I see. Yeah, you want to meet. We have to present you the, the other the other one. We are, you know,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 Euh, Περιμένουμε την άφηξη του κυρίου Τούρμες. Σύντομο διάλειμμα λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε στα ε, θέματα φαρμακευτικής Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Τύρμες που τον περιμένουμε τουλάχιστον πέντε λεπτά έφτασε. Έχουμε την κάρτα σου εδώ, Κλοντ. Θέλουμε να έρθεις εδώ μπροστά. Um, uh, Κύριε Τύρμες, ε, βρίσκεστε εδώ και ε, θα μιλήσουμε για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης. Ε, η κυρία Παρμανόβα είναι εδώ, ο κύριος Φόξ όχι. Και ο κύριος Αλπίνη. Έχουμε εδώ μεγάλη ομάδα σκιωδών εισηγητών που θα σας ακούσει. Κλοντ, ε, εν να τα συζητήσουμε τα θέματα σήμερα. Πέντε λεπτά άργησες, αλλά δεν πειράζει. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Θέλουμε λοιπόν να μας ενημερώσεις για την πολλή δουλειά που έχεις κάνει στα θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης. Ε, ήμουνα στο κέντρο με το ποδήλατό μου και ε, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσει παράνομα μέτρα για να έρθω στην ώρα μου, αλλά δεν το έκανα. Λοιπόν, θα, σας ε, κάνω μια γρήγορη εισαγωγή. Να υποθέσω ότι θα έχετε διαβάσει τη γνωμοδότησή μου. Ε, όπως είχα ανακοινώσει, βρισκόμαστε στην ΙΜΚΟ, οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα τα σημαντικά για μας, τα πυρηνικά για μας. Και γι' αυτό δεν έχω καλύψει ένα τόσο ευρύ φάσμα όσο η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η ΕΝΒΗ. Θέλω αυξημένο ρόλο για τις οργανώσεις ασθενών. Ε, ξέρουμε ότι μάλλον υπάρχουν ε, χρόνια ελλειπή στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ε, ενέργειες και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα με την εισαγωγή των ασθενών στο σύστημα. Ένα πρόβλημα με τους ασθενείς είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι ειδικοί. Οπότε όταν νιώθουν ότι ένα φάρμακο έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, θα το περιγράψουν αυτό και, με, και θα το ε, μπερδέψουν με πολλά ε, προσωπικά αισθήματα τα οποία δεν βασίζονται στην επιστήμη. Και γι' αυτό θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να τα αναλύει ένας φορέας που να μπορεί να κρίνει τι είναι υποκειμενικό και τι είναι αντικειμενικό όσον αφορά τις ε, ενέργειες αυτές. Βασιζόμαστε στην εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών αρχών ε, ώστε οι εθνικές αρχές να λαμβάνουν πληροφορίες από τους ασθενείς, από τα νοσοκομεία, από τους γιατρούς, από τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα είναι έτσι στη θέση να κάνουν μια εντελεχή ανάλυση και οι σχετικές πληροφορίες θα ε, εισάγονται στο ευρωπαϊκό σύστημα Udra Vigilance, το οποίο θα μας επιτρέψει να βασιστούμε στις ισχυρές εθνικές αρχές, ωστόσο όμως να έχουμε ένα πρόβλημα ένα, ένα σύστημα ε, που να επιτρέπει το μοίρασμα των πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εμένα με ενδιέφερε ακριβώς αυτό. Αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ελληπών στοιχείων για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα το, το πρόβλημα πώς θα διαχειριστούμε όλες τις πληροφορίες αυτές και πώς θα ξεχωρίσουμε τις ε, σημαντικές από τις μη σημαντικές. Το άλλο θέμα για το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες και για τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και για τους καταναλωτές να συμβουλεύονται δηλαδή την βάση δεδομένων Udra Vigilance Νομίζω ότι σχεδόν έχω ε, ολοκληρώσει το θέμα αυτό και θα έχετε προσέξει ότι έχω διαγράψει ένα ή δύο σημεία του κειμένου της Κομισιόν που πιστεύω ότι μάλλον θα αποδυναμώσουν την θέση των καταναλωτών, των ασθενών και την ασφάλεια των φαρμάκων. Οι γρήγορες διαδικασίες, αυτές οι διαδικασίες fast track, υπάρχουν για φάρμακα ε, που είναι απαραίτητα, όπως τα φάρμακα κατά του ιού του AIDS. Δεν θέλουμε όμως να διευρύνουμε αυτή την πρακτική υπερβολικά και το άλλο θέμα είναι η ιδέα της Κομισιόν να γίνονται περιλήψεις που ήδη οι περιλήψεις που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά φυλάδια για τα φάρμακα δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα. Θέλουμε να δώσουμε εντολή στην Κομισιόν ώστε να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα ε, των ε, φίλων αυτών για τους ασθενείς, να είναι πιο ευνόητα. Διότι εάν συμπιέσουμε υπερβολικά τις πληροφορίες, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες χρήσιμες πληροφορίες να παραληφθούν. Αυτά αυτή τη στιγμή περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή και τις προτάσεις για τροπολογίες. Ο κ. Φόξ είναι εδώ. Θα ακούσουμε όλους τους κοιόδης. Και αν κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής θέλει να μπει στον κατάλογο των ομιλητών, να κάνει ένα νεύμα προς τον κύριο Νταν. Καταρχάς, η Μπερναντέρ Βενιού έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τούρμες για την έκθεσή του που την υποδέχομαι θετικά διότι τροποποίησε πολλά σημεία της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρούσα ενδεχομένως προβληματικά. Στην οδηγία σημείωσε και θετικά στοιχεία. Υπάρχει μια σαφής βούληση για βελτίωση της διαφάνειας των πληροφοριών όσον αφορά την εποπτεία όσον αφορά τα φάρμακα, το φαρμακευτικό σύστημα και να γίνει αποτελεσματικό και πιο εύκολο να αντιδρά. Είμαι υπέρ της ενθαρρύνσεως της διαβίβασης των πληροφοριών στους ε, ασθενείς χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν στο γιατρό και να ε, τον συμβουλευτούν. Να δίδονται οι πληροφορίες από τη στιγμή που πληροφορίες αυτές διέρχονται από περιφερειακά και εθνικά κέντρα που μπορούν να διηθήσουν τις πληροφορίες. Διότι θεωρώ ότι μια άμεση επαφή με τους ασθενείς ίσως δημιουργήσει προβλήματα λόγω ποσότητας στοιχείων όσον αφορά του ελέγχου στον τομέα αυτό Χρειάζεται χρόνος ανάλυσης των στοιχείων και αν υπάρχουν πολλά στοιχεία επέρχεται μείωση της διαφάνειας. Η πρόταση ε, μια σύνοψη όσον αφορά ε, την σύνοψη των πληροφοριών που είδε στα φάρμακα διαγράφεται, κάτι που θεωρώ απαραίτητα. Μια σύνοψη δεν είναι πάντα χρήσιμη και μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο να μην γνωρίζει πλήρως ασθενής όλες τις πληροφορίες που χορηγούνται. Ε, παραμένουν και κάποιες λεπτομέρειες προς ρύθμιση και κάποια σημεία που χρειάζονται ανάλυση και προσπάθεια συμφωνίας μεταξύ μας. Όσον αφορά τη νέα διαδικασία αδειοδότησης όρους άρθρο 21α, ε, δεν θεωρώ αναγκαίο να διαγραφεί, αλλά να πλαισιωθεί διευκρινίζοντας ότι εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να παραμείνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να μην γίνει ο κανόνας. Είμαι υπέρ επίσης χρηματοδοτήσεως από το δημόσιο τομέα. Δεν είμαι κλειστή εντελώς όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω εισφορών, αλλά είναι σημαντικό να μην υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των φορέων και της φαρμακοβιομηχανίας. Θα πρέπει να αποφευχθεί η φαρμακοβιομηχανία να είναι ταυτόχρονα και δικαστής και κρινόμενος και να συμμετέχει. Λοιπόν, το διοικητικό δεν, ε, τα μέτρα για την ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα δεν μου φαίνονται επαρκή. Πρέπει να αλλάχθουν και άλλες στοιχείες που δεν αναφέρθηκαν. Χρειάζεται ανάλυση η ε, δομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ περίπλοκη και δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην εξασφάλιση ανεξαρτησία όσον αφορά την Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των φαρμάκων και την υπηρεσία που αδειοδοτεί τη διάθεση στην αγορά των φαρμάκων. Ε, και διαρωτώ με όσον αφορά την παρουσία των 27 κρατών μελών σε αυτό το νέο φορέα. Δεν ξέρω αν θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα και πρέπει να αποφύγουμε το ότι οι ασθενείς να μπορούν να δίνουν πληροφορίες απευθείας στα εργαστήρια να, να μην κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές όλα τα στοιχεία και όσον αφορά τα φάρμακα. Τα, τα ανώνυμα τα φάρμακα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν τα άλλα φάρμακα. Δεν θα πρέπει ε, να γίνεται επεξεργασία, μια ιδιαίτερη εξαίρεση. Διότι είναι φάρμακα. Δεν θα πρέπει να περνά από διαδικασία, αυτά τα ορφανά φάρμακα να περνά από μια διαδικασία πιο ε, ε, ταχεία από ό,τι τα άλλα τα κανονικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παβανόβα είναι η επόμενη. Και μετά ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και υπάρχει προφανής ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα ελέγχου των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές και ε, χαίρομαι πολύ που προτείνεται αυτή η έκθεση και να συγχαρώ τον κύριο Τούρμες για την προσπάθεια που έκανε όσον αφορά την διαφάνεια και το, αυτά που αναφέρει το φυλάδι ενημέρωση του ασθενού. Συμφωνώ με τι προτάσεις του όσον αφορά το φυλάδι αυτό, όσον αφορά τις συνοπτικές πληροφορίες, τι βασικές πληροφορίες που θα παρέχονται στου ασθενεί και τους ε, καταναλωτέ και οι διάφορες ε, οργανώσεις καταναλωτών και ασθενών συμφωνούμε την ιδέα για την ειδική προειδοποίηση ε, για ε, τα παρακολουθούμενα προϊόντα, ελεγχόμενα προϊόντα. Το τρίγωνο αυτό, το μαύρο τρίγωνο, το σύμβολο αυτό θα πρέπει ίσως να αποφευθεί γιατί μπορεί να δημιουργεί σύγχυση και να ανησυχεί τους ασθενείς και ίσως να μην πετυχαίνει αυτό που θέλουμε εμείς σαν αποτέλεσμα να ε, εφιστούμε την προσοχή του ασθενούς. θα μπορούσαμε ε, να γίνονται μελέτες μετά την αδειοδότηση. Να αναφέρεται ότι να αναφέρε, όταν βρίσκονται παρενέργειες αφού διατεθεί να προϊόν στην αγορά να μπορεί να αναφέρεται αυτό και αντί να λέμε εντατικά παρακολουθούμενα προϊόντα να χρησιμοποιήσουμε η ποιότερη έκφραση όπως προϊόντα και ο έλεγχος αυτών μετά την αδειοδότησή τους. Ίσως ε, πρέπει να αποφύγουμε τη σύγχυσα. Μην θεωρηθεί ότι δεν παρακολουθούνται επαρκώς. Οι ασθενεί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην οπτική έκθεση και πλήρης έκθεση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε επιστημονικούς φορείς γιατί αυτές οι εκθέσεις πολλές φορές έχουν χιλιάδες σελίδε και ίσως τελικά δημιουργούν σύγχυση. Και ίσως... Ε, επηρεάζουν την άποψη του ασθενού. Κάποιε εκθέσει αρκετά μακροσκελεί, εμπεριέχουν τεχνικού όρου. Οι πλήρε εκθέσει θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για έρευνα και επιστημονικού σκοπού. Όσον αφορά για το ρόλο του ΤΡΑΚ και τη μεταρρύθμιση του, του συστήματος, πρέπει να δούμε τι γίνεται μεταξύ CNHP και PRAC, κυρίως σε περιπτώσεις διαφωνιών ο εισηγητής προτείνει το πράκ να ηγείται και να αποφασίζει. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμούν να συμμετέχουν και δύο επιτροπές. Για μας είναι ανοιχτό ποια είναι η συνέπεια συνεχών διαφωνιών μεταξύ των δύο επιτροπών. Όταν μιλάμε για δημόσιες ακροάσεις θα πρέπει να επικρατεί διαφάνεια όσον αφορά το σύστημα ελέγχου των φαρμάκων και τα μέλη του CNHP μπορούν να συναντώνται με μέλη του ΤΡΑΚ για να διαργανώνονται οι δημόσιες ακροάσεις, για να καλύπτεται ευρύ φάσμα. Ανησυχώ για την αλλαγή προτείνει ο Για το στόχο η ευρωπαϊκός έλεγχος φαρμάκων να γίνει αποτελεσματικότερος. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνονται όταν εντοπίζονται αρνητικές συνέπειες στο κέντρο συλλογής αυτών των πληροφοριών για την επαγρύπνηση. Θα πρέπει οι ασθενείς να μπορούν να αναφέρουν κάποια φαινόμενα βάση δεδομένων. Πρέπει να, είναι, να, έχει πρόσβαση και αυτός που είναι κάτοχος της αδείας στη βάση δεδομένων. Σας ευχαριστώ κυρία Παβάνοβα. Ο κύριος Φόξ επόμενος και ο κύριος Ζουβέ μετά. Και θα είμαι ο τελευταίος από τους Σκιώδης. Ο κύριος Φόξ έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τούρμς για τη δουλειά που έκανε. Πρότεινε πολλές βελτιώσεις. Μπορούμε να τις στηρίξουμε. Χαιρόμαστε που υπευλήθησαν τροπολογίες που βελτιώνουν την προστασία των δεδομένων και των καταναλωτών και νομίζουμε ότι η σύναψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν παραπλανητική και ίσω τελικά οδηγεί σε αύξηση των παρεξηγήσεων όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα. Υποστηρίζουμε τη διαγραφή τη αν λόγω αναφορά από την πρόταση. Επίση, υποστηρίζουμε και τη διαγραφή του μαύρου τριγώνου. Ε, υποστηρίζουμε τον κύριο Τούρμες όσον αφορά το ότι οι εθνικές αρχές που συντονίζουν τη συλλογή στοιχείων και θα πρέπει να καταχωρούν τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές αρχές είναι οι καλύτερες για τη συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητες για να βελτιώσουν τον επαγρύπνηση των φάρμακα, τον έλεγχο των φαρμάκων. Δεν πιστεύουμε ότι η υποβολή αναφορών για τις ε, πληροφοριών πρέπει να βασίζεται μόνο στο διαδίκτυο. Δεν έχουν όλοι οι καταναλωτές πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται και να ενθαρρύνονται όλες οι μορφές επικοινωνίας για περαιτέρω βελτίωση. Αυτές οι θύρε στο διαδίκτυο των Εθνικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ενώσεω θα πρέπει να παρουσιάσουν φυλάδια με ε, ιστορικό αλλαγής ετικετοθεσίας ε, να, να βλέπουν οι κατανοτές και να κατανοούν και θα πρέπει να διατίθεται δημοσία ε, το εγχειρίδιο που είναι στη συσκευασία όταν χορηγείται η άδεια και να δίδει πλήρης ακριβείς πληροφορίες σε όλους τους καταναλωτές. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Ο κύριος Ζουβά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και και εγώ για την εκθεσή του τον κύριο Τούρμες, παρόλο που δεν συμφωνώ με όλα όσα γράφει. Μερικά πολύ σημαντικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάποια σημεία που ακούσαμε. Πρώτα απ' όλα για το συνοπτικό κείμενο όσον αφορά τις κύριες πληροφορίες, δηλαδή για το φάρμακο. Κοιτάξτε, έτσι καλώς σε σύνοψη των χαρακτηριστικών τη ουσία είναι ήδη μια περίληψη. Αν, κάνουμε, αν συνοψίσουμε την περίληψη, έπειτα τα τρία αστεράκια στο τρίγωνο μου θυμίζει, πρόεδρε, όταν στο πανεπιστήμιο δεν είχαμε ένα μαύρο τρίγωνο, αλλά είχαμε μια νεκροκεφαλή πάνω σε ένα μπουκάλι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε στα νοσοκομεία ασθενεί και οι συγγενείς τους όταν μπαίναμε με ένα τέτοιο μπουκάλι στα δωμάτια πώς ε, αντιδρούσανε. Δεν προσφέρει τίποτα. Το να λέμε φάρμακο υπό επαγρύπνηση πάλι δεν ξέρω είναι καλή ιδέα γιατί στο κάτω-κάτω όλα τα φάρμακα πρέπει να βρίσκονται υπό επαγρύπνηση. Δεν βλέπω γιατί μερικά και μερικά αλλά όχι. Ο ορισμός τώρα των ανεπιθύμητων ε, ενεργειών. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε διεθνώς με κάποιες προδιαγραφές. Για το θέμα τώρα της κοινοποίησης των ανεπιθύμητων ε, ενεργειών είναι το στοιχείο κλειδί του κειμένου. Γιατί? Γιατί μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης είναι για να αποφεύγονται τα ατυχήματα, τα οποία δεν δηλώνονται αρκετά. Και όσο δεν θα δηλώνονται όλα τα ατυχήματα από τα φάρμακα, η φάρμακοεπακρύπνηση δεν θα μπορεί να ανταποκρίνεται στο στόχο της, στον τελικό. Άρα πρέπει να υπάρχει καλύτερη δήλωση των περιπτώσεων. Πώς δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά για παράδειγμα μπορούμε να αφήνουμε στον ασθενή την ελευθερία να δηλώνει το πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έθεσε και ο συνάδελφος ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να κατακλειστούμε από δηλώσεις που δεν έχουν νόημα. Οι ασθενείς μπορούν να μας βοηθάνε για τα αρνητικά, αλλά όχι για ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με παρενέργειες. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι πολύ θετικό στην έκθεση, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Η ενία δήλωση για τις ανεπιθύμητες παρενέργειες, ναι, Προκειμένου να απλοποιήσουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε συγκέντρωση των δεδομένων. Η δήλωση, άπαξ και γίνεται από την υπηρεσία φαρμακοεπαγρύπνησης, πρέπει να υπάρχει και ένα feedback από τα κράτη-μέλη. Αν μη τι άλλο, να έχουν τις ίδιες πληροφορίες. Είναι στην πράξη πώς θα το χειριστούμε πιο πολύ και όχι θεωρία που με ενοχλεί εδώ. Πάντως πιστεύω ότι θα είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Τώρα έρχομαι στη χρηματοδότηση. Μεγάλη συζήτηση εδώ. Σα ζητάμε για το φύλλο των αγγέλων. Ορισμένοι λένε ναι, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι εντελώ από το κράτο. Άλλοι λένε η ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει να επιτρέπεται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πραγματιστέ. Να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Όλε οι δημόσιε δομέ, τη μία την άλλη στιγμή, έχουν ιδιωτική χρηματοδότηση, αν μη τι άλλο, μέσω των φόρων. Και τι λέει το κείμενο της Κομισιόν, που εγώ το βρίσκω αρκετά ισορροπημένο. Λέει, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι δημόσια, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσουμε να υπάρχουν εισφορές οι οποίες πληρώνονται από τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Από τη στιγμή λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε εκεί η κυρία Βερνιό, υπάρχει ανεξαρτησία για την χρήση των πόρων και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το δημόσιο, να είμαστε πραγματιστές, να χρησιμοποιούμε ιδιωτικά κονδύλια. Αλλά η χρήση αυτή να είναι ανεξάρτητη από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις εταιρείε. Απλά είναι τα πράγματα για μένα. Η οργάνωση δημοσίων ακροάσεων για να ξεκινήσει η κοινωτική διαδικασία έχει να κάνει με τη διαφάνεια και την ενημέρωση. Πολύ ενδιαφέρον. Η οργάνωση επίσης δημόσιο τομέα και κεφάλαια. Εδώ πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε μετά από τις ακροάσεις αυτές να υπάρξει μια πρώτη έκθεση. Να μην περιμένουμε 80 μέρες γιατί μέσα σε 80 αυτές μέρες μπορεί να ξεκινήσουν διάφορες πολεμικές που να μην έχουν ένα όνομα. Η Food Administration έχει ένα σύστημα που αμέσως έχουμε μια πρώτη έκθεση με το που τελειώνει η ακρόαση. Οπότε έχουμε μια γενική εικόνα και η κανονική έκθεση έρχεται αργότερα. Για την κατάργηση του PSUR. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι εταιρείε πρέπει περιοδικά να δίνουν κάποια έκθεση για την χρήση, τακτικά, σε τακτικό επίπεδο και προβλέπει οδηγεί, ότι κάποια φάρμακα που έχουν άδεια προκαιρού περίπου 8 χρόνια αναφέρονται. Ε, το ψήρ λοιπόν δεν είναι απαραίτητο. Μπερδεύομαι όσον αφορά αυτή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι έχουμε παραδείγματα φαρμάκων που είναι στη αγορά χρόνια και κάποια μέρα λέμε ότι πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά. Έχουν παράδειγμα στη Γαλλία ένα φάρμακο που θα αποσυρθεί οφείλονται κάποιοι θάνατοι. Για... Είναι ένα φάρμακο για... η ε, θάνατοι ήταν από νεφρική ανεπάρκεια. Και αυτό το φάρμακο που φταίει για αυτούς τους θανάτους ήταν 35-40 χρόνια στην αγορά. Ισχύει λοιπόν, είναι σημαντικό το θέμα και για τα παλιά φάρμακα. Είναι ένα κείμενο καλό, αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χρειάζεται βελτίωση ίσως γιατί δεν λειτουργεί η φάρμακοεπαγρύπνηση, δεν λειτουργεί γιατί δεν γίνεται επαρκή δήλωση περιστατικών και θα πρέπει να βελτιωθεί αυτός ο τομέας. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έδινα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να μιλήσετε πριν ή μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Στέμπεργκερ νομίζω είναι εδώ. Σύντομος παρακαλώ, γιατί έχουμε μείνει πίσω χρονικά Μετά θα δώσω και το λόγο στον κύριο Τούρμες και να επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τροπολογιών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος διότι στην παλαιότερη συζήτηση στην Επιτροπή μου δώσατε ήδη την ευκαιρία να απαντήσω σε κάποια από τα θέματα που εθίγησαν και δεν θέλω να το επαναλάβω. Θα ήθελα να τονίσω όμως δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα για την χρηματοδότηση από το δημόσιο τομέα. Να επαναλάβω ότι κατά παρελθόν η χρηματοδότηση για τη φαρμακοεπαγρύπνηση δεν αρκούσε για να αναβαθμιστεί το σύστημα στα αναγκαία επίπεδα. Είναι μια καλή ιδέα η δημόσια χρηματοδότηση. Να δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει οξύ κίνδυνος. Η ανεξαρτησία της υπηρεσίας υπονομεύεται από αυτές τις εισφορές. Διότι η υπηρεσία εν γέννη χρηματοδοτείται κατά 75% από εισφορές. Από εισφορές από την αδειοδότηση για διάθεση στην αγορά. 25% περίπου προέρχεται από κοινοτικούς ε, πόρους. Η Δημοσιονομική Αρχή εγκρίνει τα κονδύλια αυτά. Δεν αρκούν υπό αυτές τις περιστάσεις να καλύψουν τα πάντα που προβλέπει η νομοθεσία. Η αλφανά φάρμακα εξαίρεση από εισφορές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μακρύς ο κατάλογος. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λάβει υπόψη και την πραγματικότητα. δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται τα πάντα από δημόσιους πόρους. Όσον αφορά το τη φαρμακοεπαγρύπνησης, εκεί μπορεί να αποφασίσει ο φορέας μαζί με τους ε, ε, ειδικούς των κρατών μελών να κινηθεί και είναι ανεξάρτητη. Και αν στα ετήσια τέλη, σε αιτήσεις φορές συμπεριληφθεί φαρμακοεπαγρύπνηση, θα διατηρηθεί η ε, ανεξαρτησία τους. Δεν χρειάζεται ειδικό τέλος, ειδική σφορά για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Δεν δικαιολογούνται σχετικά με το θέμα οι αμφιβολίε σας. Δεύτερη αμφιβολία που έχετε είναι για την υπό όρους αδειοδότησης εξαιρετικές περιστάσεις, το περίφημο άρθρο 24α που θα θέλατε να διαγραφεί. Το έφερε κάποιος ομιλητή ότι ήδη έχουμε νομικές διατάξεις περί εξαιρετικών περιστάσεων και αδειοδότηση υπό όρους. Υπάρχει πλαισίωση και μπορεί να είναι κάποιοι όροι για μια σπάνια ασθένεια. Για να υπάρχει αναγκαίος αριθμός δοκιμών για κλινικές αποδείξεις, χρειάζεται τόσος χρόνος για κλινικές δοκιμές που δεν δικαιολογείται. Ένα παράδειγμα δίνω. Δεν θέλω να μπω τώρα σε θέματα όπως η γρήπη των πτηνών λοιπά, την πρόσφατη πανδημία και λοιπά. Εν γέννη όμως ίσως υπάρχουν περιστάσεις για να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποίησαμε συχνά αυτή τη διάταξη, αλλά μόνο σε καλά δικαιολογημένες περιστάσεις. Δεν προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γενικεύσει αυτή την προσέγγιση. Αυτή την ιδέα έχετε, αλλά δεν ανήκει στα κίνητρά μας κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να γενικευτεί αυτή η προσέγγιση. Διευκρινίζουμε, μπορεί να δοθεί αδειοδότηση υπό όρους. Και αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί με ε, μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας μετά την αδειοδότηση. Δεν αλλάζουμε τα σύνορα και λέμε ότι πρέπει να δίδονται πιο γρήγορα οι άδειε. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Δεν ξέρω πού προέρχεται αυτή η παρεξήγηση, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε εργαλεία για να πιέσουμε τη φαρμακοβιομηχανία σε ορισμένε περιστάσεις να δώσει στοιχεία και να αυξηθεί η επαγρύπνηση και ο έλεγχος σε ειδικέ περιστάσεις. Αυτό θέλαμε να το ξεκαθαρίσουμε και νομίζω ότι έχουμε καλούς λόγους για κάτι τέτοιο. Παρακαλώ δεχτείτε την εξήγησή μου. Δεν έχουμε κάποιες κρυμμένες προθέσεις σε αυτή την περίπτωση. Και τέλος, είμαστε υπέρ προστασίας δεδομένων και με το Συμβούλιο συζητούμε πώς μπορούμε να βασιστούμε στην γνωμοδότηση για τον Ευρωπαίο επόπτη των στοιχείων. Όσον αφορά το φυλάδιο της συσκευασία και για την σύνοψη, ακούστηκαν και θετικά σχόλια και είδα ποιο είναι το μήνυμα και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ότι αυτή η ιδέα δεν βρίσκει πολλούς υποστηρικτές Οπότε αυτό θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Κλοντ Τούρμες για να συνοψίσει αν το επιθυμεί και να ε, μας συνοψίσει το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση της Επιτροπής. Έχει αναφερθεί αλλού ότι εάν δώσουμε τη δυνατότητα για πιο γρήγορη έγκριση υπό κάποιες συνθήκες αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Αφού υπήρχε τόσο λίγη ανάγκη για κάτι τέτοιο στο παρελθόν, γιατί θα το χρειαστούμε στο μέλλον. Φαίνεται ότι το παρόν σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις ε, που εμφανίζονται. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Ε, στη συζήτηση σήμερα είδαμε σε ποιου τομεί υπάρχει ευρεία συνένεση και σε ποια σημεία χρειάζεται μια πιο αναλυτική ρύθμιση. Εάν όλοι δέχεστε ότι πρέπει οι ασθενεί να έχουν καλύτερες δυνατότητες συμμετοχής, τότε το βασικό θέμα είναι καλύτερο είναι να έχουμε εθνικά φίλτρα, εθνικά και περιφερειακά φίλτρα, τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, δηλαδή προτού τα στοιχεία ε, εισαχθούν στο σύστημα Ultra Vigilance. Εγώ φοβάμαι ότι εάν όλα τα δεδομένα αυτά παρακάμψουν τα εθνικά συστήματα. Δεν ξέρω πώς εργάζονται στο Vigilance, αλλά οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να επιλογή των, ε, αληθινών, των πραγματικών στοιχείων και δεν ξέρω πόσοι εργάζονται στη Vigilance, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε για χιλιάδες. Θα πρόκειται Λοιπόν, για σημαντικό λάθος κατά τη γνώμη μου, να μην επωφεληθούμε από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη, διότι εκεί βρίσκεται, ε, εκεί έχουμε πολλή γνώση και θα πρέπει να συζητήσουμε τα εθνικά συστήματα είναι αρκετά καλά ώστε κατόπιν να εισάγονται οι πληροφορίες στο ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι η προστιθέμενη αξία παράλληλα να στέλνονται τα στοιχεία στη Vigilance, διότι ε, θα κατακλειστεί το σύστημα αυτό όπως αναφέρατε και αν δεν έχουμε αρκετούς υπαλλήλου ε, που να εργάζονται στο Vigilance, τότε θα κολλήσει το σύστημα, θα υπάρξει συμφόρηση. Εγώ θέλω το επίπεδο αυτό να είναι το επίπεδο όπου ε, διανέμονται οι πληροφορίες που ήδη έχουν περάσει από κάποια φίλτρα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε εδώ αν μπορούμε να καταφέρουμε να να έχουμε συνένεση και όταν περάσει και η προθεσμία των τροπολογιών να δούμε μήπως μπορούμε να επιδιώξουμε κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, κύριε Πρόεδρε, το αφήνω σε εσά. Ε, ζητώ και πάλι συγγνώμη που άργησα. Θα προσπαθήσω να δώσω καλύτερο παράδειγμα την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολλή δουλειά που έχεις κάνει. Ευχαριστώ και τους εσκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι έχεις πολύ καλή γνώση του θέματος αυτού. Χρειάζεται να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα διότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι στη δική μας Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 23 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες που προτείνουμε είναι 2 Φεβρουαρίου την επόμενη εβδομάδα ώστε να έχουμε χρόνο να τις εξετάσουμε και εξέταση των τροπολογιών και ψηφοφορία θα πρέπει να γίνει την ίδια μέρα αλλά είμαι βέβαιος ότι θα θέλεις να συνεργαστείς με τους κοιόδης συζητητές πριν από αυτό. Ε, λυπάμαι για το περιοριστικό χρονοδιάγραμμα αλλά ε, βρισκόμαστε υποποίηση και ε, τον Απρίλιο θα πάει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Η ημερομηνία για τους κοιόδες είναι το μεσημέρι της Δευτέρας Φεβρουαρίου. Ε, ευχαριστώ πολύ Κλωτήρμες για τη δουλειά σου αυτή και να προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα στον τομέα των φαρμάκων της κυρίας Μπάστος, την οποία καλωσορίζω. Πρόκειται για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Έχουμε σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Μπάστος και θα την παρακαλούσα να μας την παρουσιάσει. Ε, να δω ποιοι είναι εδώ από τους ε, η κυρία Βάιλερ Παρβάλοβα, ο κύριος Φόξ, ε, ο κύριος Αντεγκάρτ δεν είναι εδώ. Ε, Σερβίν δεν είναι εδώ. Να υποθέσω ότι είναι κάποιος παρόν και από την Επιτροπή. Κύριε Τζέρκαρτ, θα απαντήσετε και εσείς, ε, θα απαντήσετε εσείς και σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Στέρμπεργκερ είναι υπεύθυνο από την Επιτροπή. Ωραία. Ε, ζητώ συγγνώμη, έχουμε καθυστερήσει λίγο. Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Μπάστος ε, θα καλύψει περιληπτικά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω όντω να είμαι σύντομη. Αυτή είναι μια πρόταση οδηγίας, πολύ σημαντική όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια της προστασίας των καταναλωτών. Πρόκειται για την ε, αλυσίδα διαμονής φαρμάκων, τα οποία είναι απομίμηση φαρμάκων ουσιαστικά. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα όπω ονομάζονται. Έχουν υπάρξει πολλές συναντήσεις με όλε τις εμπλεκόμενε πλευρές, με όλου τους φορείς, έχουν γίνει ερωτήσει στην Κομισιόν, συναντήσεις με τους ηγητέ, τους κοιόδης, ακροάσει. και μία μόνο διαπιστώσαμε ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Χρειάστηκε να επικεντρωθούμε και σε άλλες πτυχές που θα συμπεριλαμβάνονταν εδώ. Επίσης είχαμε και μία άτυπη συνάντηση με την Μαρία Ματίας, με την Τερέσα Πίντο επίσης που είναι βοηθός από το ΕΛΚ και όλους τους συνεργάτες αυτούς θέλω να τους ευχαριστήσω. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης απορρέει από μια ανταλλαγή απόψεων που ξεκίνησε εδώ στην Επιτροπή μας όπου εντοπίστηκαν κάποια από τα σημεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ελλειπή θέλαμε να τα διευκρινίσουμε περισσότερο. Αυτά τα σημεία λοιπόν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο γνωμοδότησής μου, στην αιτιολογική σκέψη. Εκεί μιλάω κυρίως για την ανάγκη που υπάρχει να καθορίσουμε το τι είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Τα προϊόντα αυτά τα έχουμε κυρίως μέσω ίντερνετ, μέσω διαδικτύου. Η Κομισιόν όμως δεν μιλάει για την εμπορία μέσω διαδικτύου. Εμείς γι' αυτό κάνουμε μια σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου τα επόμενα χρόνια να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις επιπτώσεις από τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην οδηγία. Ξέρουμε επίση ότι είναι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δίνουν την άδεια για την πώληση μέσω διαδικτύου των προϊόντων αυτών ή όχι. Τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα. Τα φάρμακα αυτά ως επιτοπλίστων πολλούνται μέσω διαδικτύου όμως. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να συλλέξουμε πληροφορίες από τους καταναλωτέ και να προχωρήσουμε σε αναρμόνιση των μέτρων τα οποία εφαρμόζονται και επίσης να έχουμε και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για το φαινόμενο αυτό της απομίμησης φαρμάκων. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές και απέναντι στις νέες διατάξεις ε, προστασίας. Μια άλλη πτυχή που μας ενδιαφέρει πολύ είναι ότι έχει να κάνει με τις νέες διατάξεις ακριβώς αυτές ασφάλειας. Εφαρμόζονται χρειάζεται κάποια συνταγή ιατρική, αλλά προσοχή να μην μπερδεύουμε τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται συνταγή ιατρική με εκείνα για τα οποία δεν απαιτείται τέτοια συνταγή. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Επιτροπή σε δύο χρόνια πρέπει να έχει παρουσιάσει μια έκθεση για την πραγματικότητα που ισχύει για τα φάρμακα εκείνα τα οποία ε, δεν ε, ε, τα παίρνει ο ασθενή μόνο με ιατρική συνταγή, αλλά πολλούνται ελεύθερα. Μια άλλη πτυχή έχει να κάνει με τις πληροφορίες που έχουμε βάσει κοινοτικών δεδομένων. Θα έπρεπε να υπάρχουν για να μπορούμε να εντοπίζουμε τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε την περίπτωση ε, τέτοιων φαρμάκων που έχουμε βρει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαχείριση της βάσης αυτής δεδομένων ε, πρέπει να είναι στα χέρια ειδικών αρχών των κρατών μελών. Αρχών που πρέπει να ενημερώνουν την τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση καταρχήν σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια να υπάρχει συντονισμός από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων, από τον εντοπισμό μέχρι την παρακολούθηση, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την νομοθεσία ισχύει στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά δεν θα πρέπει να είναι στη διάθεση ε, άλλων για εμπορικού σκοπούς. Όχι, γι' αυτό ακριβώς και αυτό γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι η απομίμηση φαρμάκων είναι ένα έγκλημα. Οργανωμένο πολλές φορές. Και γι' αυτό και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αποτρεπτικών μέτρων και κυρώσεων. Δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθορίσει πλαίσιο κυρώσεων, Γι' αυτό και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις δικές τους διατάξεις που έχουν να κάνουν με κυρώσεις σε αυτή την περίπτωση. Τέλος, με την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, εφαρμόζονται νέες διατάξεις, νέοι κανόνες από 1 Δεκεμβρίου του 2009. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησής μου. Όμως να προσθέσω κάτι τελευταίο. Έχοντας διαβάσει το σχέδιο γνωμοδότησης που συνέταξα με τη βοήθεια των συνεργατών και διαφόρων αρχών που σας ανέφερα στην αρχή, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο αυτό σε ορισμένα σημεία έχει κάποιες ελλείψεις λόγω μετάφρασης ή λόγω δομής. Κάποια σημεία δηλαδή πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα για να έχουμε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα στο κείμενο. Γι' αυτό και θα ήθελα στη δικιά μου τη γνωμοδότηση να υποβάλω τροπολογίες μέσα στα πλαίσια ε, τις προθεσμίες για κατάθεση τροπολογιών με στόχο τη διασφάλιση της αφήνειας, της ασφάλειας για ορισμένα σημεία που πιστεύω ότι δεν διευκρινίζονται παρκώς στο κείμενο. Είμαι στη διάθεσή σας τώρα. Ό,τι απόψεις έχετε, σχόλια, ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πάστος εάν μπορούμε από τους κοιόδες ηγητές να έχουμε επίσης περιληπτικές παρεμβάσεις. Έχω την κυρία Βάιλερ, την κυρία Παρμανόβα και τον κύριο Φόξ μέχρι στιγμής. Ε, υπάρχει άλλος που θέλει το λόγο. Η κυρία Βάιλερ πρώτη. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, σίγουρα. Λίγες παρατηρήσεις έχω. Καταρχήν, διάβασα την έκθεσή σας μόνο στα αγγλικά, όχι στα γερμανικά. Δεν υπάρχουν ακόμα οι μεταφράσεις, δεν είναι τραγικό αυτό. Δέκα τροπολογίες ε, μπορώ να τις ε, εξετάσω στα αγγλικά. Αλλά Εάν θέλουμε τροπολογίες μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, τότε θα λιγοστέψει ο χρόνος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, παραμένει η ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου, διότι τότε δεν θα προλάβουμε πολλά. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτη ερώτηση. Ε, μπορεί να μπορώ να βρω την απάντηση στην έκθεσή τη ΕΝΒΙ, αλλά ίσω μπορείτε και εσεί να μου το πείτε. Τι στόχο έχει η βάση δεδομένων αυτή. Λέτε ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίε ε, θα πρέπει να εισάγονται στη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων, λέτε, θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρεί τα κριτήρια για την προστασία των δεδομένων και να μην χρησιμοποιείται για άλλους οικονομικούς στόχους. Και αυτό είναι λογικό. Τι στόχο έχει η βάση δεδομένων. Θα πρόκειται για μια μυστική βάση δεδομένων που θα ε, βρίσκεται στη διάθεση μόνο κάποιων εμπειρογνωμόνων ε, για τα φάρμακα, ε, διότι στην περίπτωση αυτή θα έχει μόνο ένα στόχο. Θα πρέπει να είναι σαφές. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά πλαστά φάρμακα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ε, τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται. Ε, τώρα συχνά ε, τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται κατά τύχη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από γιατρούς στον οποίο τα χέρια πέφτουν τα φάρμακα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της δημοκρατίας μας, τέτοια τέτοιες εγκληματικές πράξεις, όπως λέτε πολύ σωστά, να δημοσιεύονται. Και αυτό όσον αφορά τη βάση δεδομένων. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Στις εξηγήσεις σας, περιγράφεται αρκετά αναλυτικά την συμπερίληψη των ε, αγορών μέσω διαδικτύου στην ε, οδηγία αλλά στο μεταξύ βλέπω να μιλάμε για over the counter, OTC, ε, στο κατάστημα. Αυτό δεν γίνεται μέσω διαδικτύου. Ε, μπορείτε παρακαλώ να μου αναφέρετε πού έχετε συμπεριλάβει τις επιγραμμικές πωλήσει και αν όχι ε, να υποβάλω εγώ σχετική τροπολογία. Τώρα έτσι γρήγορα που κοίταξα δεν βρήκα το σχετικό σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παρβανόβα. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μπάστος για την έκθεση. Συνεργάστηκε τέλεια, έλαβε υπόψη όλες τις προτάσεις μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τις διευκρινήσεις. Ο ορισμός των ψευτοφαρμάκων, παρόλο που μπορούμε να προσθέσουμε ότι κάθε στοιχείο του ορισμού μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά, ενίσχυση των ποινικών κυρώσεων κατά εκείνων που φτιάχνουν τα ψεύτικα φάρμακα και θα πρέπει όλοι οι και να τιμωρούνται και όλοι όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα διανομής αυτών είναι πολύ καλό. Αυτό δίνει προστιθέμενη εξή, ειδικά μέσα για την ενημέρωση των καταναλωτών για την πώληση διαδικτύου, ευαισθητοποίηση για τις πωλήσει φαρμάκων στο διαδικτύο. Η κυρία Ματία στην Επιτροπή Περιβάλλοντα έκανε έξοχη δουλειά και προτείνει κάποια πράγματα. Να υπάρχει σύστημα πιστοποίησεως των φαρμακείων των ηλεκτρονικών, των εικονικών να ενισχυθεί συνεργασία και κατάρτιση για τους τελωνιακούς και εκθέσει αξιολόγηση στην εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας δύο χρόνια μετά την εκτέλεση των μέτρων, την υλοποίηση των μέτρων από πλευρά ΣΥΜΚΟ. Υποστηρίζουμε αυτή τη γνωμοδότηση με κάποια στοιχεία που αφορούν την οργάνωση εταιρικής αγοράς και προστασία των καταναλωτών. Η ε, εκ νέου συσκευασία, η ανασυσκευασία δεν το θέτει η κυρία Μπάστο στην έκθεσή της ο καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι δεν είναι ψεύτικα τα φάρμακα είναι τα φάρμακα που έχουν ασφαλή χαρακτηριστικά. Το πακέτο συσκευασία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του προϊόντος. Τα φάρμακα δεν είναι απλά αγαθά, σαν γιαούρτι, τηλεοπτική συσκευή ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω όμως τι είναι αυτό που μπαίνει σε μια συσκευασία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως την ασφάλεια των πολιτών και την υγεία τους. Για τα γενικά φάρμακα και τις πωλήσει επιτόπου over the counter, λιγότερο από 1% των γενικών αυτών φαρμάκων, των ανωνύμων φαρμάκων παραπιούνται. Και η προσέγγιση για τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την τιμή του φαρμάκου για τις πωλήσει over the counter. Έχουμε πρώτες εκθέσεις για προϊόντα τα οποία παραποιούνται σε μεγάλο βαθμό μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και διάταξη τη Μπάστο σχετικά με τι ποινικέ κυρώσει. Για περίπτωση κατασκευή παρασκευή ψευτοφαρμάκων. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των αρχών, των αστυνομικών, των δικαστικών, τελωνιακών για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα αυτό, η παραγωγή ψευτοφαρμάκων και μία ακόμη φορά θα θέλατε συγχαρώ που έλαβε υπόψη όλες τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Μπάστος για την έκθεσή της, την γνωμοδότησή της. Είναι λογική, ε, απαντάει καλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα μας αρέσει η ρήτρα. Εμείς θα θέλαμε μετά από πέντε χρόνια, μετά τη θέση σε ισχύ, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και ορισμός των παραπημένων προϊόντων και ευχαριστούμε την κυρία Μπάστο για το έργο της επ' αυτού. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ως καταναλωτές και θα ήθελα τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης για μέτρα ασφάλειας. Ιδιαίτερα για τους κινδύνους από την αγορά φαρμάκων μέσω διαδικτύου από χώρους που δεν είναι επιστοποιημένοι. Η ομάδα μου δεν πιστεύει ότι πρώτος αυτή πρέπει να συμπεριλάβει διατάξεις για κυρώσεις, ποινικέ κυρώσεις. Αυτό είναι θέμα κρατών μελών, πιστεύουμε. Θέλουμε να εξετάσουμε περισσότερο τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ μας. Στο μεταξύ θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μια μελέτη αξιολόγησης, να δούμε τι στοιχεία θα συλλεχθούν τελικά όσον αφορά την σκοπιμότητα τη σχέση κέρδους-κόστους. Να δούμε επίσης σε εθνικό επίπεδο τι συστήματα ισχύουν και πώς έχει διανομή στην κάθε χώρα. Γιατί η κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα διανομής. Τέλος, θέλουμε όσοι ασχολούνται με το παράλληλο εμπόριο να δίνουν στοιχεία εγγύσεων. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Κύριε Τέρπεγκο. Α, συγγνώμη, ο κύριος Σβάμπ πρώτα. Θέλετε οπωσδήποτε το λόγο. Ναι. Τότε, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό όμως. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια για αυτή τη γνωμοδότηση που είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ καλή και θέλω να αποφελθώ από την ευκαιρία αυτή που εξετάζουμε τα ψευδεπίγραφα φάρμακα για να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα φόρουμ το οποίο οργανώνεται και έχει να κάνει με την πειρατεία προϊόντων. Το Μάρτιο θα λάβει χώρα συνάντηση αυτή η διάσκεψη που θα συμπεριλάβει και τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Γι' αυτό και σας καλώ να συνεισφέρετε και να συμμετάσχετε στη διάσκεψη αυτή. Ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας καλέσω στη διάσκεψη αυτή που θα λάβει η χώρα το Μάρτιο, όπως σας είπα. Ωραία, τώρα κύριο Στέρβαγκερ. Πολύ σύντομο όμως, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Μία παρατήρηση για τις κυρώσεις. Γίνονται διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης για ποινικέ κυρώσεις για παραπημένα φάρμακα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν προχωρήσει πολύ. Βέβαια, η Κομισιόν έχει στηρίξει αυτές τις διαπραγματεύσεις και πολιτικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Αλλά είναι ένα νομικό ζήτημα που ιδίω μετά από αυτά που είπε ο κ. Φόξ ήθελα να το θέσω. Για τη βάση δεδομένων τώρα και για περιπτώσεις μέσα σε μια βάση δεδομένων και αυτό συζητήθηκε. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, υπάρχει σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών δηλαδή μεταξύ των κρατών μελών και πρόθεση είναι η δημιουργία μια ειδική ανταλλαγή ε, απόψεων μέσω των εθνικών αρμοδίων υπηρεσιών που δεν θα είναι μια βάση δεδομένων αλλά θα είναι μια ανταλλαγή απόψεων προωθημένη για τα φάρμακα αυτά. Έπειτα, και το καθεστώς έχουμε πει και στο παρελθόν ότι θα ήταν μια ιδέα για την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων ε, μέσω διαδικτύου. Η ενημέρωση των καταναλωτών είναι όντως περιορισμένη σήμερα, πρέπει να ενισχυθεί. Γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με νέες προτάσεις από πλευρά της Επιτροπής και να δούμε χρειάζεται περισσότερο μια νομοθετική ρύθμιση, χρειάζονται περισσότερο πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν ξέρουμε. Για να καταπολεμήσουμε επίσης την πώληση ψευδεπίγραφων φαρμάκων ε, μέσω διαδικτύου ή μέσω παράνομων δικτύων. Για την ε, μελέτη σκοπιμότητας δεν νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να περισσότερο σε βάθος να πάμε. Η Επιτροπή ΕΝΒΗ θα το δει αυτό πιο πολύ. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πάντως ένα εμπορικό απόρριτο εδώ. Αν υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες, καλό θα ήταν να μην υπάρξει κατάχρηση των δεδομένων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Θα πρέπει να καλύπτονται από το απόρριτο. Έτσι εμείς καταλαβαίνουμε την πρόθεση αυτή που υπάρχει. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπάστος τώρα. Θέλετε να συνοψίσετε. Έχω και ένα χρονοδιάγραμμα για να ανακοινώσω, οπότε σύντομα παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Μπάστος. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τα σχόλιά τους. Πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά. Έτσι θα μπορέσω να συνεχίσω με την προετοιμασία της γνωμοδότησης αυτής συνοπτικά, πρέπει να σας πω ότι για τις ανησυχίες της κυρίας Βάιλερ, όσον αφορά τη βάση δεδομένων, βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπάντησε και είπε ότι η βάση αυτή δεδομένων υπήρχε ήδη για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και ότι τώρα πρέπει να υπάρξει μια ειδική βάση δεδομένων για την απομίμηση φαρμάκων. Για τις διατάξεις ασφάλειας τώρα και το εμπορικό απόρριτο δεν είναι πράγματα τα οποία ε, μπορούν να δημοσιευθούν. Γιατί ακριβώ πρέπει να τηρούν το απόρριτο. Όσο για το διαδίκτυο θα θέλαμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Είναι εξάλλου μία από τις επικρίσεις που είχαμε για αυτήν την πρόταση. Είναι μια πρόταση οδηγίας που μπαίνει στην αλυσίδα των ε, νόμιμων φαρμάκων καταρχήν και για την δυνατότητα πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, νόμιμα πολλούνται φάρμακα μέσω διαδικτύου, ενώ σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν ή να δίνουν άδειε για τέτοιου είδους πώληση φαρμάκων δηλαδή μέσω διαδικτύου. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο της παραποίησης φαρμάκων γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου. Επειδή όμως δεν αναφέρεται σε τροπολογία ειδικά, γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προβλέψει μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης και η Επιτροπή βλέπω ότι συμφωνεί προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τον πραγματικό κίνδυνο που ελοχεύει στην περίπτωση αγοράς φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να είναι σίγουροι ότι είναι ασφαλής η αγορά αυτή που θα κάνουν. Τώρα για το ερώτημα της κυρίας Παρμανόβα για τις ετικέτες των μπουκαλιών. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που προσπαθήσαμε να εξετάσουμε στην έκθεση. Υπάρχει ανησυχία για την προέλευση των φαρμάκων, για να βρούμε τα ίχνη των φαρμάκων αυτών, αν υπάρχει παράλληλο εμπόριο για τα φάρμακα. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι φορείς της αλυσίδας πρέπει να μοιράζονται την ίδια ευθύνη. Έχουν όλοι ευθύνη. Αυτό το παράλληλο εμπόριο λοιπόν πρέπει να έχει τις ίδιες ευθύνες όπως έχουν και οι άλλοι φορείς. Πρέπει να υιοθετούν αντίστοιχες διατάξεις και να έχουν την υποχρέωση εγγύησης όσον αφορά την προέλευση του φαρμάκου. Αν υπάρχει αυτή η εγγύηση, εντάξει. Δεν μπορούμε αυτή την εγγύηση να την αφήσουμε απ' έξω. Είναι μια οικονομική πραγματικότητα. Στον τομέα των φαρμάκων. Αυτό το παράλληλο εμπόριο. Ναι, ναι. Πρόεδρος διακόπτη, πρέπει να σας ζητήσω να ολοκληρώσετε. Η κυρία Μπάστος, ναι, ναι, εντάξει, τελείωσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, ήθελα να ολοκληρώσετε στα γρήγορα. Αν θέλετε να περάσετε κάποια σημαντικά μηνύματα στο τέλος, καλώς. Να ανακοινώσω τη σπάση, το χρονοδιάγραμμα, το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα. Ψηφοφορία στην καθήλια αρμόδια επιτροπή τον Απρίλιο προτείνουμε προθεσμία για τροπολογίες 9 Φεβρουαρίου για τους κοιόδης έξετας τροπολογιών 16 Μαρτίου και θα ψηφίσουμε στις 17 Μαρτίου. Συμφωνείτε κυρία Μπάστος. Ωραία. Θα υπάρξει και άλλη ευκαιρία να διεξαχθεί συζήτηση επί των τροπολογιών και μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποια άλλα σημεία. Και ζητώ συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά έχουμε πολλά άλλα σημεία να εξετάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Τώρα θα προχωρήσουμε. Νέα προγράμματα που ξεκινάνε σήμερα. Ζητώ συγγνώμη από τον Λουί Γκρέκ που είναι ο μεθεπόμενος και τον Φραντσεσκόφσκι, αλλά έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και έχουμε πολλά να εξετάσουμε. Παρακαλώ και τους δύο να σκιαγραφίσουν τι έχουν υπόψη τους όσον αφορά το πεδίο που θα καλύπτει η έκθεση και σκιώδεις μπορούν να σχολιάσουν σύντομα σχετικά ζητήματα και ας μην μπουν στην ουσία διότι την ουσία θα έχουμε την ευκαιρία στα πλαίσια της εκθέσεως να τη συζητήσουμε. Έκθεση ιδίας πρωτοβουλία όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο Ελβετία εμπόδια όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Ο κ. Τσασκόφσκι είναι ο εισηγητής. Ο κ. Μήτρο Ρέπο είναι εδώ ο κ. Κρόιτσμαν, η κυρία Ρούλε δεν είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ, είμαι ο σκιώδης σας και Σαβίνη δεν είναι εδώ και δεν ξέρω αν επιθυμεί να σχολιάσει και κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω κυρία Ντέιλι ότι θα πάρει το λόγο τώρα, θα ακούσει αυτά που έχουμε να πούμε. Κύριε Τρασκόφσκι, μπορείτε να αναφερθείτε στο έγγραφο εργασίας σας και να μας πείτε πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε πάνω σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από λίγα λόγια για το έγγραφο εργασίας, να σκιαγραφίσω δύο επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Θα αναφερθούμε σε δύο διαφορετικά πράγματα. Χώρες που είναι μέλη της εσωτερικής αγοράς συνεργάζονται μαζί μας στενά με την εσωτερική αγορά αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και προφανώς έχουμε τον ΕΟΧ θεσμοθετημένο σύστημα, δυναμικό, σύγχρονο όπου τα μέλη του ΕΟΧ συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον αφορά την υλοποίηση και απ' την άλλη έχουμε ένα σύστημα με την Ελβετία που βασίζεται σε 120 διμερείς συμφωνίες Πολύ περίπλοκο το σύστημα με 27 μεικτέ επιτροπέ για τη λήψη αποφάσεων. Δεν υπάρχει μια ομορφή εφαρμογή κανόνων εσωτερική αγορά. Υπάρχει έλλειψη ασφαλεία δικαίου και επιστομή κλπ. Ευθύ εξ αρχή θέλαμε να εξετάσουμε και τα δύο ζητήματα. Μετά από πολλέ συζητήσει, όμω, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα με την Ελβετία και την ΕΟΧ, Ελβετία και ΕΟΧ δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα τώρα. Το έγγραφο εργασίας μας αντιμετωπίζει, εξετάζει την φύση των σχέσεων Ελβετίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αφού μίλησα μαζί σας όμως και με κάποιους άλλους συναδέλφους, αποφασίσαμε να σκεφτούμε κατά πόσο πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχική πρόταση, να εξετάσουμε το θέμα του ΕΟΧ και να έχουμε ένα έγγραφο που θα είναι πιο μακρόπνο, να εξετάσουμε θέματα όπως είναι δημοσυμβάσεις, δικαιώματα καταναλωτών κλπ. Και από ό,τι κατάλαβα συμφώνησαν οι συγγητές να επιστρέψουμε στην ευρύτερη προσέγγιση που θα καλύπτει και τον ΕΟΧ, θα οργανώνονταν και μία μήνυα κρόαση και θα είχαμε τη δυνατότητα να καλέσουμε και τους εταίρους της ΕΟΧ να συμμετάσχουν στη συζήτηση και εν τη αυτή περιπτώσει θα έπρεπε να αναβληθεί τη τελική μορφή του σχεδίου εκθέσεως γιατί χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε διότι το έγγραφο εργασίας πρωτίστως ασχολείται με την Ελβετία. Όσον αφορά το έγγραφο εργασίας, αυτό κάθε αυτό, το έχετε μπροστά σας. Θα πω μερικά λόγια γι' αυτό. Στην αρχή περιγράφει το σύστημα σχέσεων μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πολύ περίπλοκο σύστημα και δύσκολο να εξηγηθεί σε μερικές παραγράφους. Το σημαντικότερο είναι ότι είναι στατικό σύστημα και περιέχει πολλά προβλήματα, κυρίως για μας που έχουμε συνηθίσει τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά. Παράδειγμα, δεν υπάρχει άμεση συνέπεια αυτών των διατάξεων στην Ελβετία. Δεν υπάρχει ομοιόμορφη υλοποίηση και εφαρμογή και ακόμα και το δόγμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέει ότι δεν υπάρχει παράλληλη ερμηνεία. Η πρόσφατη απόφαση του 2009 Εκεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ των δύο συστημάτων. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα ακόμα. Όταν μιλάμε για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, παραδείγματο χάρη, ακρογωνίως λίθο του συστήματο τη εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, είναι η αρχή του Κασί Ντεντιζόν. Δεν ισχύει στην Ελβετία αυτή η περίφημη υπόθεση. Μετά εξαίρεση για δημόσια συμφέροντα, για την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών, εφαρμόζεται διακριτικά στην Ελβετία κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα παρεμφέρει. Υπάρχουν κάποια εμπόδια για την ελεύθερη διακίνηση ατόμων και υπηρεσιών, τα οποία αναφέρουμε στο έγγραφο εργασία και πολλά μέλη θα θέλουν να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Όπως χρειάζεται κοινοποίηση 8 ημερών, αν μιλάμε για παροχή υπηρεσιών συγγνώμη σε περισσότερα καντόνια της Ελβετίας. Αυτό δημιουργεί απλώ εμπόδιο, αλλά εφαρμόζεται με διακριτικό τρόπο γιατί ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του υπηκόου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στο τέλος του εγγράφου εργασίας θέτουμε κάποια ερωτήματα για περαιτέρω συζήτηση, διότι θέλουμε αυτό το έγγραφο να στρέφεται προς το μέλλον. Το σημαντικότερο πως να διευκολυνθεί η διευθέτηση διαφορών, διότι όπως είπα δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου στο σύστημα. Δεύτερον, πως να εξασφαλίζουμε πιο έγκαιρη σύγκληση νομοθεσίας ελβετικής που απεισέ εσωτερική αγορά, πώς θα εφαρμόσουμε τις συμφωνίες στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Και αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο διότι δεν υπάρχει γενική συμφωνία για την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εφαρμογή μιας γενικής συμφωνίας πάνω στο θέμα και το γενικότερο θέμα που θα πρέπει πιθανότατα να συζητηθεί εκτενέστερα. Κατά πόσο θα πρέπει να εστιαστούμε επιβελτιώσεως του κεκτημένου, του status quo, να βελτιώσουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων που είναι περιπλοκότατη ή να προχωρήσουμε πιο πέρα και να βάλουμε μια συμφωνία πλαίσιο που θα είναι πολύ φιλόδοξη και θα εμπεριέχει δυναμικά στοιχεία. Να υπενθυμίσω λοιπόν το βασικό δίλημα που σκιαγράφησα στην αρχή. Μπορούμε να κάνουμε τα εξή. Πρώτον, να εστιαστούμε στην Ελβετία. Προ τα εκεί πάει το έγγραφο εργασία. Δεύτερον, εναλλακτική να θετήσουμε την ευρύτερη προσέγγιση που ήθελαν περισσότεροι συνάδελφοι. Δηλαδή, θα αναφερθούμε και στον ΕΟΧ, θα αναφερθούμε σε μελλοντικά θέματα όπως είναι δικαιώματα καταναλωτών και ε, δημόσιες προμήθειες και θα χρειαζόταν μήνυ ακρόαση περισσότερος χρόνος, τα είχαμε σχέδιο εκθέσεως όχι σε μια εβδομάδα όπως ήταν αρχική πρόθεση αλλά σε ένα μήνα και οι συντονιστές πήραν αυτή την απόφαση, αλλά εσείς τελικά θα εγκρίνετε ή θα επιβεβαιώσετε αυτή την απόφαση των ε, συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή παρέμβαση αυτή και να μιλήσω και ως πρόεδρος και ως κοιόδης εισηγητής τη ομάδας μου για το θέμα αυτό και ελπίζω να συμφωνήσουν ο κύριος Ρέπο και ο κύριος Κρότσμαν. Νομίζω ότι οι συντονιστές το συζήτησαν αυτό και στην συνάντηση στρατηγική στην Τρίτη και θεώρησαν ότι θα πρέπει να είναι ευρεία η έκθεση αυτή και ήδη νωρί στη θητεία μας να καλέσουμε εκπροσώπους από τον ε, ΕΟΧ και την Ελβετία. Και θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονός ότι έχουμε ένα έγγραφο ενημέρωσης για τον ΕΟΧ και την Ελβετία. μια σχετική ενημέρωση νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη και για το χρονοδιάγραμμά σας, διότι περιλαμβάνετε πολλές χρήσιμες προτάσεις. Γενικά, πιστεύω, ότι αυτή είναι η πρόταση των συντονιστών προς την Επιτροπή, με την οποία νομίζω ότι συμφωνείτε και θα σας παρακαλούσα μαζί με τους κοιόδης να εκπονήσετε χρονοδιάγραμμα και να βρείτε και μια ημερομηνία για ακρόαση. επιτρέψτε μου να ακούσουμε σύντομα τον κύριο Ρέπο και τον κύριο Κρότσμαν, να δούμε αν συμφωνούν με την προσέγγιση αυτή, να ακούσουμε και άλλες παρατηρήσεις. Κατόπιν κύριε Τσασκόφσκι, θα σας ξαναδώσουμε το λόγο ε, για να προωθήσετε την υπόθεση. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο εργασία αυτό αποτελεί πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας. Μπορεί να μην είναι απίστευτα φιλόδοξα, καθότι είναι τα θέματα αυτά αρκετά αντικειμενικά. Ε, Θα ήθελα να ξέρω πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία να λύσουν τα μεταξύ τους προβλήματα ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται χωρίς προβλήματα. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ενδιαφέρον ερώτημα θα είναι η Ελβετία θα μετακινηθεί στι θέσει τη ή όχι. Υπάρχουν πολλέ προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας της διαπριμένης εσωτερικής αγοράς και όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι το θέμα Ελβετία και εσωτερική αγορά. Αρκεί να σκεφτούμε την ε, συζήτηση σχετικά με την αποκάλυψη των τόκων. Ε, οι Ευρωπαίοι δεν τα κατάφεραν, οι Αμερικανοί όμως με τις απειλές τους και με τις ε, ισχυρές απαιτήσει τους κατάφεραν να κινήσουν τα πράγματα. Το θέμα είναι η Ελβετία θέλει να βελτιώσει την κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτό έχει νόημα να συζητάμε για διεύρυνση στις χώρες ΕΖΕΣ. Έχω εντύπωση ότι πιο εύκολα θα προχωρήσουμε με τις χώρες ΕΖΕΣ παρά με την Ελβετία. Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ελβετία με την πολύ ισχυρή άμεση δημοκρατία της, με τα δημοψηφίσματα, έχει προβλήματα. Ωστόσο, υπάρχουν εκθέσεις, ε, αναφορές οι οποίε δεν αναγνωρίζουν πράγματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην Ελβετία. Θα προσπαθήσω να έχω συζήτηση με τους ενδιαφερομένους, ε, να δούμε σε τι βαθμό υπάρχει ε, ενδιαφέρον διμερός ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να, ε, τις χώρες ΕΖΕΣ να δημιουργηθεί, να σημειωθεί πρόοδος να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις. Για παράδειγμα, να έχουμε κοινέ επιτροπές οι οποίες ε, να ε, συναντώνται και να συζητάνε τα θέματα αυτά. Θα πρέπει καταρχήν όμως να διαπιστώσουμε αν υπάρχει η διάθεση από την άλλη πλευρά και αν υπάρχει μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σβάμπ, ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό, διότι νομίζω ότι μένετε πιο κοντά στην Ελβετία από εμά. Εν πάση περιπτώσει ότι συνορεύει με την Ελβετία η ε, ε, ε, εκλογική σα περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο, γιατί ξέρω ότι μα πιέζει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τρασκόφσκι για την πλήρη και αντικειμενική του δουλειά εκ μέρους της Επιτροπής μας. Βρίσκω ότι είναι πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας. Ε, ναι, και πράγματι είμαι γείτονας της Ελβετίας ε, και ε, επηρεάζομαι από πολλά από τα προβλήματα που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά. Μερικά δεν, ήξερα καν. ωστόσο θα πρέπει να υποθεί ότι η ίδια η Ελβετία στις διμερείς ε, σχέσεις έχει διαφορετική μεταχείριση από ότι η Νορβηγία, το Λίχτενστάιν και η Ισλανδία. Ο συνάδελφος Σταρσκόφσκι όμως είπε ότι μπορεί να το λάβει και αυτό υπόψη του. Δεύτερον θα ήθελα να πω ότι... Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά όπως είπε και ο κύριος Κρότσμαν από τους ε, φιλελευθέρους τις δυσκολίες που έχει η Ελβετία με την άμεση δημοκρατία και τη μη αναγνώριση των δικαστηρίων. Εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με πολλούς Ελβετούς συναδέρφους, ε, ωστόσο οι διμερεί ε, ε, συμφωνίε Ευρωπαϊκής Ένωση και Ελβετίας στο βαθμό που ισχύουν θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν επιτρέπονται δικαιολογίε για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν εξετάσουμε την πρόταση του κυρίου Τρασκόφσκι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε την εφαρμογή των όσων ήδη έχουν συμφωνηθεί. Και όσον αφορά ε, κάτι που θα βοηθήσει όχι μόνο τους ε, παρόχους υπηρεσιών αλλά και ε, πολλούς άλλους που εμπορεύονται με την Ελβετία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σφάπ. Κύριε Τρασκόσκη, μήπως θέλετε να συνοψίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή μας δίνει την ευκαιρία για τρία πράγματα. Καταρχήν να έχουμε μια, ένα στιγμιότυπο, μια φωτογραφία της ε, σχέσης ε, που ε, αποτελεί μια πολύ καλή σύνοψη όλων των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε. Και παρεμπιπτόντω, το έγγραφο εργασία που αναφέρετε είναι εξαιρετικό. Θα αποτελέσει πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας για θέματα της εσωτερικής αγοράς. Δεύτερον, η νέα προσέγγιση απέναντι στον ΕΟΧ μα επιτρέπει να συμμετέχουν και οι εταίροι μας. Και αυτό είναι καλό διότι έτσι δείχνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί. Η ψύχρεμη ματιά απ' έξω των δικών μας προβλημάτων ε, μπορεί συχνά να μας διαφωτίζει. Γιατί λοιπόν να μην το κάνουμε. Ε, τρίτον, ε, θέλουμε να προτείνουμε κάποιε λύσει και στα πλαίσια του status quo με την σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Μπορούμε λοιπόν να κοιτάξουμε το μέλλον και να δούμε μήπω θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο υπάρχον μορφότυπο. Ε, ευχαριστώ πολύ ε, για τις ε, παρεμβάσεις σας. Θα συνεργαστώ με τους κοιόδης εισηγητές. Θα είμαι σε στενή επαφή με τους γραμματείς. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε μια μήνυα ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σασκόφσκι. Όταν θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα θα σας το ανακοινώσουμε. Έχουμε συνεδρίαση στις 8 Φεβρουαρίου. Θα μπορέσουμε λοιπόν να σα δώσουμε ένα-δύο λεπτά να μα αναφέρετε το χρονοδιάγραμμα ώστε να γνωρίζουμε όλοι πού βρισκόμαστε. Η άλλη μου παρατήρηση είναι ότι είμαστε η Επιτροπή Εσωτερική Αγορά, όχι εξωτερικών υποθέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να επικεντρωθούμε στι στοιχείε που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά. Ήδη έχω μιλήσει με την κυρία Γόλη που είναι αντιπρόεδρο ε, ε, ε, τη αντιπροσωπεία για την Ελβετία. Οπότε καλό θα είναι να συμμετέχουμε συμμετέχουν και αυτοί. Ναι, είμαστε σε στενή επαφή και του ε, κάλεσαν να συμμετάσχουν στη συζήτησή μα. Ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε παράλληλα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και περνάμε στο επόμενο θέμα μας σήμερα. Είναι μια σημαντική έκθεση του κύριου Γκρέχ για την παράδοση μιας ενιαίας αγοράς στους καταναλωτές και τους πολίτες μας. Δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος Γκρέχ λοιπόν, παρακαλώ, να συνοψίσει τις κύριες ιδέες της έκθεσής του και μετά να μιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Να έχουμε μετά τον κύριο Κάρα, τον κύριο Ροσφόρ, εγώ, ο κύριος Διόρ επίσης και ο ηγητές. Σύντομα, παρακαλώ όλοι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα την ανταλλαγή απόψεων και θα έχουμε την ευκαιρία και άλλη φορά να συνεχίσουμε. Παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Γκρέχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε επιστολή που εστάλει στον καθηγητή Μόντι, το θέσαμε μια mission impossible. Παραμένει η εσωτερική και ενιαία μας αγορά ως λίθος για την Ευρώπη. Με αυτό συμφωνούμε όλοι. Όπως όμως όλοι επίσης ξέρουμε, η ακρογωνία η λήθη πρέπει να είναι λύθη. Που πρέπει να είναι άρα στέρεη, γερή. Η ενία αγορά λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτή είναι μια δικασία που δεν είναι αφίδρομη. Είναι μια δύσκολη διαδικασία που δεν πρέπει κανείς να θεωρεί δεδομένη. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία των καταναλωτών. Δεν είναι δεδομένη. Και θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι εδώ πέρα εφευρίσκω τον τροχό. Ε, αν έλεγα ότι καταλαβαίνω πώς λειτουργεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να επαναδιατυπώσουμε την ενιαία αγορά βάζοντας τον καταναλωτή στο κέντρο της όλης διαδικασίας προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας και την οικονομική σημερινή πραγματικότητα αλλά και τις προτεραιότητες των καταναλωτών σήμερα και στο μέλλον. Η αντίληψη των καταναλωτών όσον αφορά την ενιαία αγορά είναι συγκεχημένοι, αρνητικοί συχνά ή τη θεωρούν ανύπαρκτη. Μιλήστε με τους συμπολίτε σας και ρωτήστε τους τι είναι η προστασία του καταναλωτή σήμερα, τι είναι η αγορά. Ε, λοιπόν, πολύ συχνά θα ακούσετε μια σιωπή. Αυτό πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει αμέσως. Η πρόσφατη κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να μας ε, οδηγήσει σε αποφάσεις βιαστικές, όμως η οικονομική πραγματικότητα όντως πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αποφασίζουμε για αναζωγόνηση της ενίας αγοράς. Εγώ σκοπεύω και προτείνω στην έκθεσή μου να συμπεριλάβω τους εξής κύριους στόχους. Πρώτον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τον τελευταίο καιρό προκειμένου αυτή η ενιαία αγορά να γίνει βιώσιμη. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ποιοι είναι οι στόχοι μας ως ΙΜΚΟ και ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενιαία αγορά, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το 2012. Και τέλος πρέπει να προτείνουμε νέα μέτρα για να αντιστρέψουμε τη σημερινή κατάσταση. Προτείνω λοιπόν η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2010 να μας παρουσιάσει έγγραφο με προτάσεις για νέα νομοθετική ατζέντα όσον αφορά την ενιαία αγορά, ξεκινώντας από τους στόχους της συνθήκης, δηλαδή να πετύχουμε μια ανταγωνιστική κοινωνική και οικονομική αγορά. Μια σφαιρική λοιπόν προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τους ε, φραγμούς, την πραγματικότητα, την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Η Επιτροπή πρέπει να μας παρουσιάσει μια νέα ατζέντα για την ενία αγορά και εκεί ο καταναλωτής να βρίσκεται στην καρδιά της ενίας αγοράς. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει η συμμεταχείριση και ισορροπία μεταξύ όλων των φορέων και των εμπλεκομένων. Ένας άλλος στόχος πρέπει να είναι η προστασία του καταναλωτή αυτόματα να είναι ακρογωνίας λίθος για κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σκοπεύω να προτείνω να ασχοληθούμε με την καλύτερη νομοθετική ρύθμιση να δούμε ποιο είναι το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις και να έχουμε πιο επικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τους ρυθμιστέ και την Κομισιόν. Πρέπει να υπογραμμίζουμε στην έκθεση αυτή μια σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της τρέχουσας νομοθεσίας που παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για πολλού. Ο κύριος Μπαρνιέ το είπε στην ακρόασή του ότι πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ το θέμα της μεταφοράς της νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία. Τα εμπόδια υπάρχουν, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να έχουμε μια αποτελεσματική ενιαία αγορά και να προχωρήσει ώστε να έχει την καλύτερη δυνατόν επίδοση για όλους. Πολύ συχνά τα κράτη-μέλη δεν καταφέρουν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο ή να εφαρμόσουν σωστά την κοινοτική νομοθεσία. Και αυτό είναι σε βάρος του καταναλωτή συνήθως. Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν νιώθει, δεν νιώθουν τα κράτη-μέλη, δεν συνεργάζονται αρκετά και δεν νιώθουν δικά τους όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος, πολλές φορές λείπει η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ενή αγορά. Πρέπει να αποφύγουμε τον προστατευτισμό ή την επανεθνικοποίηση πολιτικών. Αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε συχνά και στο μέλλον. Κάποια λοιπόν από τα δικά μέτρα τα οποία θα προτείνω θα είναι καλύτερης ποιότητας νομοθεσία. Νομοθεσία και για τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Solvit, να επεκτείνουμε επίσης την ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, να αντιμετωπίσουμε την παραποίηση των προϊόντων, το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας επίσης και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της, ε, του εμπορίου online. Καλύτερες διατάξεις επίσης για διασυνοριακές υπηρεσίες. Όλα αυτά θα αποτελέσουν το πλαίσιο της εκθεσής μου. Εννοείται ότι δεν μου φαίνεται εύκολη δουλειά. Ξέρω ότι είναι η δουλειά μας και η δικιά σας και η δικιά μου να βάλουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Αυτό λοιπόν θα φροντίσω να κάνω. Προτείνω έπρεπε να έχω ένα σχέδιο έκθεσης. Θέλω όμως πρώτα να ακούσω τους σκιώδες εισηγητές Γι' αυτό να μην είναι για τις 8 του μηνός, αλλά να δώσουμε περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε όλοι όσοι θέλουν, κυρίως οι σκιώδες εισηγητές, να έχουν χρόνο για να μας μεταφέρουν τις απόψεις τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ, Λουί, λοιπόν. Και εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα, πολύ φιλόδοξο. Όπως είπα, δυστυχώς έχουμε ξεμείνει από χρόνο, διότι έχουμε και την έκθεση της κυρίας Σαρτόρη Καλό τους κοιόδης ίσως να σχολιάσουν εν συντομία τη γενική προσέγγιση χωρίς να επισέλθουμε σε αυτή τη φάση σε λεπτομέρειες. Και το χρονοδιάγραμμα, αν γίνει αυτό, θα με βοηθούσε. Ο Όθμαν, Ρόθμαν Κάρας είναι εδώ, τον καλωσορίζω στην Επιτροπή. Μετά ο κύριος Ροσφόρ. Και μετά θα κάνω... Ο κύριος Ντεγιόγκ είναι εδώ, θα του δώσω το λόγο. Και στη σύνοψη που θα κάνω θα συμπεριλάβω και τις δικές μου απόψεις. Ο Ότμαν Κάρας, ήθελα. Κύριε Πρόεδρε, πρώτη παρατήρηση. Χαίρομαι για τη συνέχιση της εργασίας ε, με τον εισηγητή. Η εσωτερική αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει μεγάλο δυναμικό και αποτελεί μία από τις απαντήσεις ε, στην οικονομική και δημοσιονομική κρίση και στην παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό θα πρέπει να εξαλείψουμε τα εμπόδια εντός της εσωτερικής αγοράς. Και δεύτερον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εσωτερική αγορά δεν αποτελεί μόνο θέμα ε, νομικών ρυθμίσεων. Είναι και θέμα επένδυσης, έρευνας, εκπαίδευσης, ε, ε, φορολογικής πολιτικής και περιφερειακής πολιτικής. Γι' αυτό θα πρέπει να καλέσουμε την Κομισιόν να υποβάλει ισολογισμό σχετικά με τις οι οικονομικές συνθήκες για ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, ποια είναι τα εμπόδια της κοινή αγοράς και θα πρέπει να ε, εκπονήσει έναν κατάλογο κριτηρίων. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι η εξής. Έχουμε τώρα την συνθήκη της Λισαβόνας που αποτελεί νέα βάση για τις εργασίες μας. Έχουμε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες και αυτό είναι ένας τρόπος να επηρεάσουμε την ε, ε, ε, πολιτική. Έχουμε την πλήρη απασχόληση σαν στόχο στη συνθήκη και έχουμε και την ανταγωνιστικότητα ως μέσο για να τα πετύχουμε αυτά. Αυτά τα σημεία αυτά θα πρέπει να παίξουν ρόλο στην διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για νέο πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχει αυτή η αντίθεση, η κοινωνική συνοχή, η οικονομική ανταγωνιστικότητα. Τρίτη μου παρατήρηση. Έχουμε λόγω των διαφορών στην ανταγωνιστικότητα προβλήματα. Χρειαζόμαστε ε, ισχυρό συντονισμό στην εφορολογική πολιτική, στην κοινωνική πολιτική, στην εκπαιδευτική πολιτική και στην πολιτική έρευνας. Εάν δεν πετύχουμε περισσότερο ευρωπαϊκό συντονισμό, δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε με τον βέλτιστο τρόπο την εσωτερική αγορά. Διότι τα θέματα της, ευρωπαϊκής, της ε, εσωτερικής αγοράς είναι ευρωπαϊκά. Έχουμε τη Small Business Act, την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε όμως την αρμοδιότητα για να την εφαρμόσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να αποτελεί αυτό μέρος ε, της όλης σύλληψης της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πώς ε, καλύπτουμε την εσωτερική αγορά παροχής υπηρεσιών ε, στην έκθεσή μας ε, για την εσωτερική αγορά. Πρόκειται για πολύ σημαντικό ερώτημα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα νέα αυτά σημεία στις εργασίες μας και να καταφέρουμε και να κινήσουμε την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριο Ροσφόρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Γκρέκ σωστά παρέθεσε όλα τα σημαντικά θέματα που τίθενται, τα ζητήματα αυτά. Που είναι πολύ σημαντικό το θέμα της αναζωγόνησης της εσωτερικής αγοράς. Να πω ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε θα ήταν θεωρήσουμε ότι είναι ευκαιρία η αποστολή του κυρίου Μόντι. Να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία που δημιουργείται από την αποστολή που θα τον θέσει ο πρόεδρος Μπαρόσο να βάλει τούρμπο στο κινητήρα στροβιλοσυμπιεστή με άλλα λόγια. Όπως είπατε λοιπόν, χρειάζεται πιο γενική προσέγγιση. Μία ανάλυση που μπαίνει στη ρίζα των προβλημάτων. Ε, ε, δημιουργείται κόποση της ενίας αγοράς και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Την επικαλείται. Συντομώ λοιπόν με κάποιες ε, προτάσεις. Θα καταλάβουμε κάτι. Τι λέει. Ότι πρέπει να να δημιουργήσουμε τα πράγματα. Δεν αφορά τη βελτίωση κάποιων διαδικασιών. Χρειάζεται εκ νέου καθορισμός. Γιατί είμαστε μαζί. Χρειάζεται ανοικοδόμηση. Το νέο σύμφωνο αποκαλεί, τη νέα συμφωνία. Και πρέπει, παρόλο που καταγόμαστε φωτικέ χώρες, λέει στις χώρες που έχουν περισσότερο, υποστηρίζουν περισσότερο την ε, κοινωνική οικονομία της αγοράς, όπως είναι Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο, ότι διστάζουν να μπουν περισσότερο στην ε, ε, ε, ενιαία αγορά και λέει και στις χώρες με ε, νοτροπία που διστάζουν να εφαρμόσουν φορολογική, φορολογικό συντονισμό και κοινωνική προσέγγιση. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά να τα συναθρήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Καλά ξαναεισάγεται, κύριε Γκρέκ τον καταναλωτή γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα. Αλλά μισθωτό επίσης να είναι ο καταναλωτής, πολίτης. Θα ήθελα να ακολουθήσουμε την προτινόμενη κατεύθυνση, να την υποστηρίξουμε, γιατί θα μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές. Ίσως αργότερα ο Μισελ Μπαρνιέ ίσως μπορεί να τα λάβει αυτά υπόψη. Ακούσαμε τον κύριο Μόντι στην Επιτροπή. Υπάρχουν και τα πρακτικά χάρη στον πρόεδρο Χάρμπορ, είχαμε και lunch, γεύμα, ανθρώπων περί τον κύριο Μόντι. Λοιπόν, είναι διαθέσιμα όλα τα πρακτικά, ακούστε τα, δείτε τα. Ίσως να είπε πιο ισχυρά πράγματα ο κ. Μόντι στην συνεδρίαση από ότι αυτά που είναι στα πρακτικά των, ε, του γεύματος. Τα πρακτικά λοιπόν αυτά που σας προανέφερα και των δύο περιστάσεων είναι χρήσιμα να τα συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας κύριε Γκρέκ. Ο κύριος Ντιγιόγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κύρια πρόκληση, μια που έχουμε λίγο χρόνο για ένα τόσο σημαντικό θέμα, δεν θέλω να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Χρειαζόμαστε ένα νέο βαθμολόγιο για τα μικρότερα, τα πιο τεχνικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Πάντως συμφωνώ με του προλαλήσατε ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να κερδίσουμε την καρδιά και το μυαλό όλων των πολιτών. Αν αυτό είναι στο κέντρο της έκθεσης, το πώς δηλαδή θα το καταφέρουμε αυτό, τότε εντάξει. Τότε θα είναι πιο αποτελεσματική η εσωτερική αγορά. Αν ξέρεις ότι καταλαβαίνει ο κόσμος και είναι υπέρ της ενιαίας αγοράς, θα βοηθήσουν να πετύχει αυτή. Ξέρω ότι δεν είναι τελική συζήτηση. Μερικά σημεία μόνο θέλω να βάλω στο τραπέζι. Να πω για πράγματα τα οποία στη χώρα μου τουλάχιστον έχουν προκαλέσει επικρίσεις όσον αφορά την έννοια της ενιαίας αγοράς. Πρώτον, μερικές φορές βλέπουμε προτάσεις της Επιτροπής ή θέλει να, για παράδειγμα, να στηριχθεί ζωολογικός κήπος σε ένα δήμο. Τελικά όμως χρειάστηκε να παραδεχτεί η Επιτροπή ότι ήταν υπερβολή και δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Στη στιγμή υπάρχει ένας μόνος ζωολογικός κήπος. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Για τις δημόσιες υπηρεσίες επίσης, για μερικές τουλάχιστον, επίσης έχουμε υπερβολές. Το παράδειγμα αυτό πήρε τεράστια δημοσιοποίηση. Τεράστιες διαστάσεις και ήταν κρίμα, έκανε ζημιά. Ο κύριος Μόντι αναφέρθηκε πάντως σε αυτό το τομέα, οπότε ελπίζω ότι θα δοθεί η πρέψα προσοχή. Για μένα Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που θέλουν σε τοπικό επίπεδο να δράσουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικές φορές με την αναρμόνιση των ε, κανόνων, και η καλή ενημέρωση είναι εδώ ένα καλό παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα για αυτούς που θέλουν να μείνουν σε τοπικό επίπεδο, αλλά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις γενικές ρυθμίσεις. Γιατί εμεί θέλουμε να ρυθμίζουμε γενικά. Οπότε πώ να απλοποιήσουμε τι ρυθμίσει που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόν. Να σχολιάσω κι εγώ και μετά ο Λουί. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ροσφόρ για το που πρέπει να εστιαστούμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι έγγραφο δράσεως για τον κύριο Μπαρνιέ και για τον κύριο Μόντι και το Συμβούλιο ενδεχομένω για τους τομεί ευθυνών μας. Παρακολούθησα τον Λουί σε αυτά που είπε. Είπε να είναι μια οικονομία τη ενιαίας αγορά πολύ ανταγωνιστική, νέο πρόγραμμα να γνωστοποιηθεί στους καταναλωτές. Διαφωνώ μαζί του προ το τέλο όμω. Αναφέρθηκε σε σειρά άλλων αξιοσημείωτων ε, τομέων όπως είναι η υγεία, καταπολέμηση παραποιημένων προϊόντων, πνευματικά δικαιώματα κλπ. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μπορεί να συζητήσουμε και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά δεν θα πρέπει να υπερφορτωθούμε. Εγώ θα επέλεγα ποιότητα και στοχευμένη προσέγγιση αντί ποσότητα. Για να δείξουμε ότι καλύπτουμε όλο το κοινοβούλιο σαν επιτροπή. Υπάρχουν άλλα έγγραφα που το δείχνουν αυτό. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Προτείνω στον εισηγητή το εξή. Το ξανασυζητούμε με τη γραμματεία και προτείνουμε ένα θεωρημένο χρονοδιάγραμμα. Και συναντώμεθα ισκιώδης και προχωρούμε μετά. Λούι, μπορείς να συνοψίσεις. Θέλω να δω αν συμφωνείς με αυτή την προσέγγιση για νέο χρονοδιαγράμμα. Και μετά προχωράμε από εκεί και πέρα. Ο Λούι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους μου για τις παρεμβάσεις τους. Προφανώς δεν πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ τεχνική η έκθεση αυτή. Αυτό έγινε σαφές από την αρχή, αλλά νομίζω ότι θα Πρέπει σε ένα βαθμό να το κάνουμε. Ε, είμαι κατά των λέξεων συνθήματα. Ε, έχουμε ένα Είμαι κατά του να έχουμε ένα στόχο και να μην αναφέρουμε τα μέσα με τα οποία σκοπεύουμε να ε, πετύχουμε το στόχο αυτόν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είμαστε υπερβολικά τεχνικοί, ούτε θα πρέπει να μην είμαστε καθόλου και επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις δικές μας συστάσεις και προτάσεις. Να απαριθμίσουμε λοιπόν κάποιους στρατηγικούς στόχους. Δεν θα πρέπει να περιγράψουμε απλά πώ περιμένουμε να πετύχουμε την ολοκλήρωση αυτή χωρί τι δικέ μα συστάσει, διότι ε, υπάρχει κίνδυνο να μα επικρίνουν ότι ε, χρησιμοποιούμε τι συνηθισμένε λέξει συνθήματα και δεν μπορούμε να τι ε, συμπληρώσουμε με συγκεκριμένε δράσει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όπως σας είπα θα προτιμούσα να ε, το παρατείνω για να έχω όσο γίνεται περισσότερες συνεισφορές από τους αδέρφους μου. Πιστεύω ότι θα είναι ε, βασική η έκθεση αυτή και δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιοριστούμε σε μια αντίδραση στην οικονομική κρίση, ούτε θα πρέπει να περιοριστούμε στη δουλειά του Μόντι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποτελέσει μέρος η δουλειά του Μόντι, αλλά να αποτελεί μια δήλωση της ΣΥΜΚΟ, της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου για το πώς θα θέλαμε να δούμε να εξελίσσεται η εσωτερική αγορά. Δεν θα πρέπει να δεσμευόμαστε από ε, έτοιμες ιδέες ή από κάποια συγκεκριμένη έκθεση. Αν μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε κύριε Πρόεδρε πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω ότι μπορώ να κλείσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ξέρω ότι είναι εδώ ο κ. Στέβιτς από την ε, Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ακούσουμε την παρέμβασή σας. Ε, πιστεύω όμως ότι θα παρακολουθήσετε στενά τις εργασίες. σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για τον ενδιαφέρον σας για τη δουλειά μας. Θα ετοιμάσουμε χρονοδιάγραμμα το οποίο θα διανύμουμε σε όλους. Και τώρα έχουμε καλύψει κάποιο μέρος του χρόνου ε, που καθυστερήσαμε, ε, όχι όμως όλων. Έχουμε μισή ώρα για δύο σημαντικές εκθέσεις. Ε, με την κυρία Σαρτόρια έχουμε τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και έφτασε και η κυρία Χέντ που δυστυχώς δεν ήταν παρούσα τη Δευτέρα. Ξέρω ότι κάποιοι από τους κοιόδες συζητητές σας θα έρθουν αργότερα. Θα ήθελα να πω στην κυρία Χέτ για να το σκεφτεί πριν φτάσουμε στην εκθεσή της ότι μόλις εξετάσαμε το μελλοντικό μας χρονοδιάγραμμα έχουμε μια βραδινή συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 8 Φεβρουαρίου για να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Μπίλαν και για να έχουμε και μια πρώτη εξέταση γνωμοδότησης της Επιτροπής ε, βιομηχανία. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και τη δική σας έκθεση στην ε, ημερήσια διάταξη της συνεδρίας αυτή. Είναι τόσο ε, μεγάλη η έκθεσή σας και τόσο σημαντική που μπορούμε να έχουμε μια προκρατική συζήτηση αλλά δεν θα έχουμε το χρόνο να την εξετάσουμε εντελεχώς λόγω της συζήτησης της κυρίας Σαρτόρη. Ε, η συνάντηση αυτή που σας λέω θα είναι στις 9 η ώρα. Αν είσαστε διαθέσιμοι, προτείνω να το κάνουμε αυτό και να ε, αλλάξουμε τις προθεσμίες για ε, τις ε, τροπολογίες. Κοιτάξτε το ημερολόγιο σας, να καλωσορίσω την κυρία Σαρτόρη και να τη συζητήσω να μας ενημερώσει για την έκθεσή της. Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη φορά για την μελέτη αντικτύπου. Παρακαλώ πείτε μας λοιπόν πού βρίσκονται οι εργασίες. Ίσως μπορώ να σας βοηθήσω και να είμαι γρήγορη πρόεδρε, διότι είμαστε στη δεύτερη ανταλλαγή απόψε. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο ήδη μπορέσαμε να συζητήσουμε. Όσον αφορά την προηγούμενη φορά, σχέση με την προηγούμενη φορά, πρόσθεσα τη συμφωνία, κατόπιν συμφωνία με τη συνάδελφο Κλάστην την κάποια άρθρα που θα εξεταστούν με τις άλλες επιτροπές σύμφωνα άρθρο 50 του ιστορικού κανονισμού. Προσθέσαμε τη συμφωνία κοινή αρμοδιότητας επί κάποιων άρθρων της προτάσεως. Τα έρθρα που συνδέονται με τις συνέπειες όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών. Άρθρα 25, παράγραφος 1, 2, 6, άρθρο 28, παράγραφος 1, 7 και 9, 10, 44 παράγραφος 1, 2, 4, 9, 47 παράγραφος 2, τα άθρα 54, 58, 62. Αυτή ήταν μια καλή συμφωνία που πέτυχα με τις συναδέλφους και από αυτόν μπορούμε ιδιαίτερως να επικεντρωθούμε. Έχουμε και άλλα σημεία, άλλα θέματα προσκάλυψη σε σχέση με τη συμφωνία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όλος αυτός ο κανονισμός βλέπετε έχει αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και όχι μόνο σε θέματα που αφορούν την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στόχοι συνθισμένοι, Η αδειοδότηση να γίνει πιο εύκολη και αξιολόγηση επίσης των ουσιών των βιοκτώνων, εναρμόνιση στο μέτρο του δυνατό της ευρωπαϊκής αγοράς και των εθνικών ρυθμιστικών προσεγγίσεων, να μειωθούν οι δαπάνες όσον αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες, να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των καταναλωτών. Πολύ συχνά εκείνων που δεν είναι ειδικοί. Αυτή είναι η στόχη που προτείνουμε και επ' αυτών βασίσαμε και τις τροπολογίες. Να προβλέπονται ανταπλουστευμένες διαδικασίες για μικρές αλλαγές, να μεριμνήσουμε να λάβουμε υπόψη το σύστημα του free riding Είναι ένα σύστημα πολύ χρήσιμο, αλλά ευρέω διαδεδομένο. Είναι πολύ χρήσιμο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Να ευθυγραμμιστούν οι διατάξει για τα βιοκτώνα με τι νομοθετικέ διατάξει που ήδη υπάρχουν, κυρίω με το REACH, για να μην υπάρχουν επικαλύψεις που δεν χρησιμεύουν σε κανέναν. Να προστατεύσουμε την επεξεργασία ευαισθήτων δεδομένων, αλλά να εξασφαλιστεί και η πρόσβαση των καταναλωτών στι πληροφορίε σύστημα ελέγχων χρειάζεται που να παρέχει εχέγγυα λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα κυρίως συνδέεται με τον κίνδυνο, σχετίζεται με τον κίνδυνο. Θα σταθώ εδώ, πιστεύω τελικά ήμουν σύντομη, ίσως από τη συζήτηση θα διαφανούν σημεία προς επεξήγηση και γι' αυτό είμαι στη διάθεση των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σατόρη που θέσατε κάποια ζητήματα και δίκιο έχετε. Έχουμε συγκεκριμένη συμφωνία που διαπραγματευτήκαμε επιτυχέστατα με την περιβάλλοντος Περιβάλλοντο και σίγουρα θα εστιαστείτε επ' αυτόν αυτό. Δεν μας αποκλείω όμω να σχολιάσουμε και άλλους τομείς. Εν τη αυτή περιπτώση θα πρέπει να πάτε και να διαπραγματευτείτε στηρίζοντας τη θέση μας έναντι τη Επιτροπή Περιβάλλοντο εκεί σε τομεί που έχουμε διεκδικήσει το δικαίωμά μα να σχολιάσουμε, θα πρέπει να δεχτούν τι τροπολογίε μα. Το συζητάτε με σκιώδη. Η κυρία Γκέπχαρτ είναι εδώ, ο κύριο Μπουζόη, ο κύριο Τούρμε απουσιάζει, ο κύριο Φόξ είναι όμω εδώ. Κυρία Γκέπχαρτ πρώτα, κύριο Μπουζόη και κύριο Φόξ. Και μετά θα επιστρέψουμε στην κυρία Σαβίνη. Έχουμε τον κύριο Σπέιτ από την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, Εστέ σύντομη παρακαλώ, διότι θα υπάρχει και άλλη δυνατότητα για συζήτηση. Στις 23 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε την έκθεση Σαρτόρ, δεν αυτή η τελική συζήτηση. Τότε θα διεξαχθεί η νέα πλήρη συζήτηση. Η Εύλιν Γκέπχαρτ πρώτη. Ελπίζω να μην πρόκειται για την ε, τελική συζήτηση. Η πρώτη είναι. Και κυρία Σαρτόρη, είναι πολύ ωραίο που έχετε διαπραγματευτεί με τη συνάδελφή σας ε, από ε, την άλλη αρμόδια επιτροπή. Πολύ γρήγορα αναφέρατε μια σειρά άρθρων. Μήπως μπορείτε να μας στείλετε τα άρθρα αυτά. Συνήθως δεν εργαζόμαστε με τον τρόπο αυτόν ναι, στην ε, Επιτροπή μας. Θα ήθελα να εξετάσω εάν και η πολιτική μου ομάδα συμφωνεί με την κατανομή αυτήν. Η Επιτροπή μας θα πρέπει επίσης να εξετάσει συνολικά το θέμα. Θα σας παρακαλούσα να δώσετε σε μένα και στους άλλους κοιόδης εισηγητές γραπτός ε, τα άρθρα αυτά για να καταλάβουμε ε, ποιο είναι το αντικείμενο της συμφωνίας. Πολύ σύντομη θα είμαι, διότι δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθος στο θέμα αυτό, αλλά όσον αφορά τα διοκτώνα, το θέμα που μας ενδιαφέρει είναι από τη μία η προστασία του καταναλωτή και από την άλλη θέματα ασφαλείας, διότι συχνά μιλάμε για πολύ δηλητηριώδεις ουσίες, ε, για δύσκολα ζητήματα και ε, θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αρκετό χρόνο ώστε να εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα. Και επίσης επιτρέψτε μου ε, να ζητήσω να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορούμε να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τι συνέπειες ε, θα έχουν οι διατάξεις ε, που θα θεσπίσουμε στον τομέα αυτών. Πρόκειται για θέμα για το οποίο χρειαζόμαστε χρόνο. Πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό θέμα, το οποίο ε, όμως πολιτικά θα έχει σημαντικές συνέπειες. Αυτά είχα να πω σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καλωσορίζω την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης και τη μείωση του διοικητικού άχθους και του κόστους, διότι έτσι παραμένουν περισσότερα χρήματα για έρευνα και έτσι εταιρείε θα δίνουν καλύτερα προϊόντα στην αγορά. Η ετικετοθεσία είναι κάτι που θεωρώ υψής της σημασίας για την προστασία του καταναλωτού και η ετικετοθεσία εγγυάται ότι πληρούνται τα κριτήρια για τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος. Η σταδιακή προσέγγιση για κεντρική διαδικασία αδειοδότησης μόνο για τα βιοκτώνα χαμηλού κινδύνου είναι κάτι που καταλαβαίνω για την ώρα. Όμως συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι στην πρώτερη συζήτηση περί ανάγκης καλύτερου ορισμού των ουσιών χαμηλού κινδύνου. Και γιατί να μην επεκταθεί η κεντρική διαδικασία σε όλα τα προϊόντα. Πιστεύω ότι οι μικροαλλαγές στο θέμα διοδότησης όπως διοικητικές αλλαγές θα πρέπει να υποφεληθούν από ταχείες διαδικασίες fast track και θα δούμε πώς θα προσθέσουν τη διαδικασία για την έρευνα. Γιατί οι διοικητικές διαδικασίες δεν μπορεί να αποτελούν φραγμό για την προώθηση της έρευνας από τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Όμως, προσέξτε και τα ανανοηλικά στα παρασιτοκτόνα. Διότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιστημονικές αβεβαιότητες για την ασφάλεια αυτών, χρήσεως αυτών. Τα ανανοηλικά λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι, θα είναι ασφαλή για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Να είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο τα βιοκτόνα και προϊόντα με τα βιοκτώνα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εντό των συνόρων είναι ασφαλή, αλλά και άλλα προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό και διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Διότι ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος, πρέπει να φροντίζουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών και να κινούμεθα προ όφελο αυτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σωστά, πολύ καλά καταφέραμε να προλάβουμε να προχωρήσουμε χρονικά. Όλοι συμφωνούν ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τα βιοκτώνα είναι πολύ περιοριστική, πολύ δαπανηρή, πολύ αναποτελεσματική και αυτή είναι μια δυνατότητα να βελτιώσουμε την κατάσταση. Η ομάδα μου θέλει η ημερομηνία αναθεώρησης να έρθει πιο κοντά. Από 2023, που είναι πολύ μακριά, και να δούμε πιο γρήγορα κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό ένα κεντρικό σύστημα. Συμφωνούμε με τον κύριο Μποζόη με αυτό που είπε. Ότι ο, ο ορισμός ο τωρινός για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου είναι πολύ στενός, έπρεπε να διευρυνθεί ούτω ώστε να περάσουν περισσότερα προϊόντα από το κεντρικό σύστημα. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, κατέχουν περίπου το 75% της αγοράς αυτής και το κόστος αναπτύξεως νέων προϊόντων είναι πάρα πολύ υψηλό. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να διορθώσει η πρόταση. Θέλουμε να παρασχεθεί και άλλη βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε πιο απλούστε διαδικασία κοινοποίηση, ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να αποφασίζουν ποιοι όροι θα πρέπει να πληρούνται. Τέλος, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κριτήρια αποκλεισμού, εξαίρεσης, ε, είναι προβληματική το να απαγορευτούν κάποια προϊόντα είναι αυθαίρετη αυτή η απόφαση και περιοριστική. Να απαγορεύονται προϊόντα που απαγορεύονται από νομοθεσία για την προστασία των φυτών δεν είναι κάτι λογικό. Τα βιοκτώνα και τα φυτοφάρμακο διαφορετική ε, προσέγγιση και δεν είναι συγκρίσιμο το κόστος. Μπορούμε να το επεξεργαστούμε αυτό με την κυρία Σαρτόρη και μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλέσω. Να καλέσω την Επιτροπή να παρέμβει πολύ σύντομα ε, πριν ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σαρτόρη και συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα που προτείναμε, κύριε Σπέτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος ότι επικροτούμε πολλές από τις παρατηρήσεις που έγιναν απόψε αναγνωρίζουμε ότι η πρόταση αυτή περιλαμβάνει μια πολύ σημαντική διάσταση που αφορά την, ευρωπαϊκή, την εσωτερική αγορά και θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες ε, εγκρίνονται τα προϊόντα αυτά. Ε, είμαστε υπέρ λοιπόν ε, της περαιτέρω απλοποίησης και της βελτίωσης της κατάστασης για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας καθησυχάσω όσον αφορά τα κριτήρια αποκλεισμού. Αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα βιοκτώνα κατά περίπτωση. Η πρόταση της Επιτροπής ορίζει σαφώς ότι μπορεί να υπάρχουν λόγοι που αφορούν τη δημόσια υγεία ε, που ε, για διατήρηση κάποιας βιοκτώνας ουσίας παρότι θεωρείται επικίνδυνη Επίση, σημειώσαμε κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι χρήσιμο να εξεταστούν περαιτέρω και επικροτούμε τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει τώρα μέχρι στιγμή γενικά. Κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα είμαστε πολύ περιορισμένοι χρονικά. Ήταν μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για μια πλήρη έκθεση στις, η συζήτηση έγινε στις 5 Νοεμβρίου που έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ζητώ συγγνώμη από τη συνάδελφο λόγω παραλήψεων απέναντί της. Απεστάλησαν σε όλες πολιτικές ομάδες. Στις 13 Νοεμβρίου απεστάλησαν οι πληροφορίες σχετικά με την συμφωνία που πετέχθη με τη συνάδελφο Κλάς. Όμως παρέλειψα να έρθω σε επαφή με τους κοιόδης εισηγητές. Δεν θα ξανασυμβεί αυτό προβλέπεται συνάντηση αμέσως μετά την αποστολή της, του κειμένου στις μεταφραστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τις απόψεις που εξέφρασαν συνάδελφοι, συμφωνώ. Επαναλαμβάνω ότι είμαι πολύ ευτυχής που συζητούμε σήμερα έναν κανονισμό με όλα αυτά που σημαίνει κάτι τέτοιο. Περνάμε από μια οδηγία σε κανονισμό Δίνουμε δηλαδή βεβαιότητα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, κάτι που επιτυγχάνουν λιγότεροι οδηγίες. Διαλέγω, διαλέξαμε τον κανονισμό, άρα κάτι που αφορά όλα τα κράτη-μέλη και που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Και αυτό είναι ήδη μεγάλο βήμα πρόοδου. Άκουσα και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνώ με τη φιλοσοφική προσέγγιση αλλά ε, υπογραμμίζω κάποια πράγματα. Την απέτηση για πλούστευση, να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την προστασία ασφαλείας του καταναλωτού, να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να προσέξουμε ιδιαίτερως την ποιότητα των προϊόντων, κυρίως των προϊόντων εκείνων που έρχονται απ' έξω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και χρειάζονται κατά την άποψή μας μία ε, βεβαιότητα για την ορθή πρακτική ε, που ακολουθείται στις χώρες εκείνες που παράγονται αυτά τα προϊόντα που εισάγουμε εμείς μετά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρτόρη. Οι συντονιστές μου είπαν να γίνει διαπραγμάτευση με ενισχυμένη συνεργασία. Το θέμα είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Η εμπορία, η αμοιβή αναγνώριση. Νόμιζα ότι το είχαμε καλύψει. Όσον αφορά πάντως το χρονοδιάγραμμα, η κυρία Σαρτόρη θα στείλει στην μετάφραση στις 2 Φεβρουαρίου το σχέδιό της. Μετά θα έχουμε συζήτηση του σχεδίου γνωμοδότησης στις 23 Φεβρουαρίου. Οπότε 1η Μαρτίου θα είναι η προθεσμή για κατάθεση τροπολογιών. 16 Μαρτίου θα τη συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε στις 17. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 26 Απριλίου θα ψηφίσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλό χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να έχουν όλοι χρόνο στη διάθεσή τους. Θα έχουμε δηλαδή τρεις-τέσσερις φορές την δυνατότητα να συζητήσουμε. Ξέρω ότι η κυρία Σαρτόρη θα ξεκινήσει τη συνεργασία με τους ισκιώδεις εισηγητές και θα φροντίσει στους ομείς εκείνους όπου έχουμε ενισχυμένη συνεργασία να έχουμε και ουσιαστικές τροπολογίες για να πάνε μετά στην ε, Ολομέλεια. Για τον κύριο Πεσό ήθελα να πω ότι τα νάνο υλικά είναι ένα θέμα για το οποίο σίγουρα θα έχετε απόψεις, αλλά αυτή είναι μια γνωμοδότηση, δεν είναι επί της ουσίας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την κυρία Σαρτόρη και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Θα έπρεπε να το είχαμε ήδη συζητήσει, αλλά δεν είχαμε εδώ την κυρία Χέντ. Τώρα την έχουμε όμως. Καλώς ήρθατε. Έχει μια πολύ καλή έκθεση και θέλω εδώ να επαναλάβω αυτό που είπα και νωρίτερα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, προτείνω να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα και την τελική ψηφοφορία, αλλά να αλλάξουμε λιγάκι το χρόνο που θα έχετε για συζήτηση με τους σκιώδες συζητητές για τις 8 Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω αν μπορείτε. Αν συμφωνείτε, εντάξει. Πάντως, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την εξαίρετη έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ πολύ σύντομη. Ιδιαίτερα για τους διερμηνείς, λέει η ομιλήτρια, επειδή πρέπει να ε, κλείσουμε στις 6.30. Καταρχήν, συγγνώμη που δεν μπορούσα να είμαι εδώ ε, Δευτέρα απόγευμα είχα κολλήσει στο αεροδρόμιο της περιοχής μου στη Σουηδία. Δυστυχώς ε, αυτό συμβαίνει με τα μικρά αεροδρόμια. Δεν είχα λοιπόν ε, την ευκαιρία να έρθω εγκαίρως. Έχετε την πρόταση εκθεσής μου για την προστασία των καταναλωτών και των πίνακα αποτελεσμάτων, το scoreboard. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία μέχρι τώρα, ιδιαίτερα την ε, γραμματεία, τους σκιώδεις εισηγητές, ε, τους συνεργάτες μου αρμοδιότητά μας ε, είναι όχι μόνο να εποπτεύουμε την ε, εσωτερική αγορά, αλλά να ε, εποπτεύουμε και τα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές. Και ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές αποτελεί πολύ, καλό εργαλείο εποπτείας της αγοράς. Είναι δεύτερη φορά που συζητάμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου Ελπίζω λοιπόν να ε, συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα αυτό πολλά χρόνια στο μέλλον. Η έκθεσή μου περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων για το πώ μπορούμε να αναπτύξουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων, νέου δείκτε, χρηματοδότηση, συλλογή στοιχείων, εποπτεία τη αγορά, ολοκλήρωση τη αγορά, ε, πρόσβαση σε ένδικα μέσα, καθώ και προτάσει ε, για το πώ η εποπτεία και οι καταναλωτικοί κανόνε μπορούν να βελτιωθούν. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πω σε περισσότερες λεπτομέρειε, διότι δεν έχουμε πολύ ε, χρόνο. Ε, θα προτιμούσα να ακούσω τι έχουν να πούν οι σκιώδεις εισηγητές και ο Πρόεδρος. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, ώστε ε, στις 2 Φεβρουαρίου στι 12 να μπορέσουμε να έχουμε την προθεσμία. Δυστυχώς μένω σε περιοχή της Σουηδίας με μικρό αεροδρόμιο και δεν προλαβαίνω να βρίσκομαι στο Στρασβούργο Δευτέρα 9 η ώρα. Ε, υποθέτω ότι θα έχουμε ε, συνάντηση των σκιωδών εισηγητών όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, μετά την ε, παραλαβή των τροπολογιών για να δούμε αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα κλείσω εδώ. Καλώς. Ούτε σκιώδες δεν έχουμε τέτοια ώρα. Ωραία, ο κύριος Μότη δεν είναι εδώ. Η κυρία Κρέμη. Α, είσαστε εκεί. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε την παρέμβαση. Δεν σας είχα δει, αν ήσασταν εδώ. Ε, τώρα εκεί πίσω που έχετε πάει και έχετε καθίσει. Η κυρία Κόμη λοιπόν εδώ για τον κύριο Μότη. Του είναι δεν εδώ, εγώ είμαι εδώ. Ούτε ο είναι εδώ. Καλά, κύριε ακόμη από το υπερπέραν. Για πείτε μας τα σχόλιά σας και ο Πίτερ Μέιερ είναι εδώ. Ιδού, στην τελευταία σειρά, όπως έκανα στο σχολείο. Επιστρέφω λοιπόν στο παρελθόν. Λοιπόν, ο κύριος Μότι μου άφησε κάποια σημεία. Πρώτα απ' όλα απευθύνει συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια για την έξοχη δουλειά της και έχει κάποιες προτάσεις και κάποιες σκέψεις. Το πρώτο αφορά την αξιοπιστία του πλαίσιου αξιολόγησης. Πιστεύει το πλαίσιο αξιολόγησης των καταναλωτών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά ακόμα πάρα πολύ ατελές. Τα στοιχεία που δίδονται από τα κράτη-μέλη, που δεν δόθηκαν ακόμα και μερικά, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είναι μη ομοιογενούς τυπολογίας, άρα δύσκολο να μπορέσουν να ομοδοποιηθούν τα στοιχεία αυτά. Ο κύριο Μότι πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να ερμηνεύουμε βιαστικά τα στοιχεία τα οποία είναι ατελή. Δεύτερον, ισορροπία μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών. Οι καταναλωτές μόνοι τους ή ομοδοποιημένοι έχουν περισσότερα μέσα στη διαθεσή τους μέσω των οποίων μπορούν να πετύχουν ορατότητα και να κρίνουν μαζικά. Θα πρέπει να πετύχουμε ισορροπία όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών και τα δικαιώματα και καθήκοντα του παραγωγού το να μιλάμε για δημιουργία υπηρεσιών καταναλωτών με πλήρες εξουσίες όπως αναφέρει το σημείο 38 της εκθέσεως θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλεισίματα αντί να οδηγήσει σε ανοίγματα, σε δημοκρατικό διάλογο που είναι ε, βάση της νομοθεσίας μας. Κάτι σημαντικό είναι εναλλακτικέ μέθοδος διευθετήσεως των διαφορών Ίσως διότι η μεσολάβηση και συμφιλίωση και άλλη μέθοδο επιλύσεως διαφορών, εξοδικαστικές μέθοδοι, είναι πάρα πολύ σημαντικά μέσα και εν αυτή περιπτώσει λιγότερα επαχθεί για τους ε, καταναλωτές, για τους πολίτες μάλλον. Θα θέλαμε να συναντηθεί και Μότι με την ε, εισηγήτρια ε, να συζητηθούν κάποια σημεία. Πρέπει να οριστεί η ενεργός πολιτική για τους καταναλωτές, στο σημείο 4 μετά, όσον αφορά το πώς υποστηρίζονται οι οργανώσεις των καταναλωτών, ε, δεν υπάρχουν διευκρινήσεις. Στο σημείο 7 προβλέπεται στα σχολαστικά προγράμματα από την παιδική ηλικία η εκπαίδευση για την κατανάλωση. Και τελευταίο σημείο, θα εκτιμάται η καλή αναλογία που προβλέπεται στο σημείο 32, όμως θα πρέπει ίσως να καταβληθεί και άλλη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη να δώσουν και άλλα χρήματα. Τέτοια εποχή ε, οικονομικής κρίσης για εντατική πολιτική για να γίνει καλύτερη αξιολόγηση και να καλύπτει ευρύτερο πεδίο και ταυτόχρονα πιστεύει ότι το θεσμικό επίπεδο και το μη κυβερνητικό επίπεδο ήδη είναι ένα επίπεδο όπου υπάρχουν οι φορείς που έχουν επομιστεί να ενημερώνουν δεόντως τα, ε, τους πολίτες για δικαιώματα τους. Άφησα τις σημειώσει ο κ. Νότι ευχαριστώντας την εισηγήτρια και εκφράζει τη λύπη για την απουσία του. Πρόεδρε, κύριε Χέντ, θα γίνεται πιο σύντομος. Με παρατηρήσεις με στόχο να βελτιώσουν την ε, κατά τα λεξαίρετη έκθεσή σας. Πρώτον, η υπεράσπιση του scoreboard, του βαθμολογίου. Είναι πολύ σημαντικό. Και το λέω γιατί από ό,τι κατάλαβα όσον αφορά την τροφοδότηση δεδομένων τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Φταίει ο συντονισμός ανάμεσα στις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίε και την Eurostat, τα είναι υπηρεσίε της Κομισιόν, δεν ξέρω. Είναι δύσκολη η συνεργασία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρώπου ιδιαίτερα υψηλού τεχνολογικού επίπεδου. Δεν είμαστε εμεί που θα καταλήξουμε στο ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο, αλλά τα διάφορα Ινστιτούτα θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται για να έχουμε αξιόπιστε πληροφορίε. Δεύτερον, τα μέσα που έχουν οι ανεξάρτητε υπηρεσίε. Εδώ δεν συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητε υπηρεσίε που να στηρίζουν τον καταναλωτή, που να τον προστατεύουν, που να μην είναι ψεύτο υπηρεσίε και να μην ε, κινδυνεύουν ε, οι οργανώσεις των καταναλωτών. Η λογική πρέπει να είναι λογική διαλόγου. Στη Γαλλία πάνε σχετικά καλά τα πράγματα. Οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι παρούσες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα ήταν να τις είχαμε όμως. Κάποια στιγμή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε για την ιδέα μιας αντίστοιχης ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Τρίτον, για τα θέματα κατάρτισης. Μιλάτε για την ενημέρωση και την κατάρτιση του καταναλωτή. Στο σχολείο λέτε εσείς. Για μένα δεν είναι μόνο στο σχολείο, είναι διαβίου και αφορά όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Αυτοί που είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση εξαιτία της οικονομικής κρίσης είναι ακριβώς αυτοί που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση για την κατανάλωση. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο υπερβολικής κατανάλωση. Πολλέ φορέ δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τη διάκριση του τι είναι χρήσιμο και τι όχι. Τέλο, Δεν είμαι πεπισμένος γιατί στο σημείο 44 μιλάτε για την εποπτεία των αγορών και μιλάτε για την δυνατότητα στιγματισμού της μιας ή της άλλης επιχείρησης θεωρώντα ότι θα ήταν καλύτερο να ξέρει ο καταναλωτή κάθε φορά ποια εταιρεία φταίει. Δεν λέω ότι είμαι εντελώ κατά μια τέτοια αρχής. Θα μπορούσε ίσως να αιτιολογείται για κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις και όταν υπάρχουν συνεχώς προβλήματα. Αλλά το να καταδεικνύουμε αμέσω όταν πρόκειται για μικρές κυρίως επιχειρήσεις αυτό καταλαβαίνετε ότι τις δυσκολεύει πολύ γρήγορα αν στιγματιστούν και οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για αυτές. Ξέρετε ότι όταν μας βάζουν στο ειδόλιο τα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και αν αποδειχτεί μετά ότι έχει γίνει λάθος, άντε να αποκατασταθεί η τιμή αυτού που έχει μπει στο ειδόλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω με μια τροπολογία, μάλλον με πολλές τροπολογίες, να ε, σας ζητήσω να λάβετε υπόψη σας τις θέσεις μου αυτές. Ο κύριος Χάρμπορ. Ευχαριστώ κύριο Φόρημος, και ο συγητής για την ομάδα μου και συμμερίζουμε την άποψή σε αυτή την έκθεση. Είναι πάρα πολύ περιεκτική και συγχαίρω την Άννα γιατί συμπεριλαμβάνει τόσα πράγματα και γι' αυτό νομίζω ότι θα την αδικήσουμε σήμερα το απόγευμα. Την αδικούμε μάλλον και ελπίζω να την πείσουμε να είναι και στο Στρασβούργο αγκαίρος για να τη συζητήσουμε εκτενέστερα τα βασικά θέματα που έχω να θίξω. Είναι θέματα γενικής αντίληψης, γενικότερα. Τι μας λένε όλα αυτά τα στοιχεία, Φερρυπίν. Καλά λέει ότι υπάρχει περιθώριο βελτιώσεως των στοιχείων και έχει σχετικώς ιδέες και για επέκταση του πεδίου που καλύπτουν. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πολιτικό του μανιφέστο αναφέρει Φέρεται σε πρωτοβουλία ελέγχου παρακολούθησης τη αγορά για πιο συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ολοκλήρωση της ενιαία αγοράς. Ίσως να αναφέρεται σε αυτό, ίσως πρέπει να το ψάξουμε. Μπορεί να μα διαφορτήσει του ο κ. Μάιρ. Αυτό σχετίζεται με τη δουλειά του Λουί Γκρέκ, όπου εκεί αναφερόμαστε στο scoreboard, στο σύστημα βαθμολόγηση εσωτερική αγορά και θέλαμε κάποιους δείκτες να τους συναθρήσουμε σε ένα πιο δομημένο τρόπο, σύστημα. Πρέπει να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προβληματικές αγορές, θα μας βοηθούσε αυτό. Ψάξατε και βρήκατε τη σημασία ε, γενικής έρευνας για τις αγορές τι ε, τις ε, στο διαδίκτυο που δείχνει τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τις ψηφιακές αγορές. Ε, ποια θα είναι η μελλοντική στρατηγική, ποιος θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που θα συλλέγονται. Τέλικα, ένα στρατηγικό θέμα. Κάτι που είναι προαπαιτούμενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η έρευνα και η καινοτομία. Τα στοιχεία για νέα προϊόντα και αναδυόμενες υπηρεσίες, κυρίως το διαδίκτυο και σε άλλους τομείς είναι σημαντικότατα στοιχεία. Ενθαρρύνουν επιτυχείς καινοτομίες και βοηθούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τους δίνουν ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικό όταν γνωρίζουν η μία τι κάνει η άλλη, τις καινοτομίες. Ίσως μπορεί να είναι ευρύτερο το πλαίσιο σαν αυτά τα στοιχεία αντί να παρακολουθούμε απλώς το πώς λειτουργεί η αγορά. Να δούμε πώς συνδέονται αυτά με τους στόχους. Ε, οικονομική ανανέωση, καινοτομία, ασφάλεια προϊόντων, όλα αυτά μπορούν να μπουν μαζί. Οπότε σίγουρα θα υποβάλουμε σχετικώ τροπολογίε. Προσβλέπουμε στην δυνατότητα να συναντηθούμε και να αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτά τα ζητήματα. Να σα ξαναδώσω το λόγο ή να αναφέρω το χρονοδιάγραμμα πριν πάρει το λόγο. Χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, τι προτείνουμε. Προθεσμία για τροπολογίε 2 Φεβρουαρίου την επόμενη εβδομάδα και αν συμφωνείτε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων εκτενέστερη 8 Φεβρουαρίου 8 Φεβρουαρίου 9 και 4 το βράδυ Στρασβούργο 21 και 15 συζήτηση 20 Φεβρουαρίου των τροπολογιών ψηφοφορία στις 23 Φεβρουαρίου την ίδια μέρα για να μπει στην ε, Ολομέλεια του Μαρτίου. Η καλύτερη προσφορά είναι αυτή φοβούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ήταν αρκετά σαφές αυτό, αλλά μπορούμε να συναντηθούμε στο αεροδρόμιο στο Στρασβούργο στις 9 και 4 άμα θέλετε. Είναι η μόνη μου δυνατότητα να φτάσω στο Στρασβούργο. 9 η ώρα το βράδυ είναι η άφηξή μου. Θα φτάσω στο Κοινοβούλιο όσο μπορώ πιο γρήγορα, αλλά... Αλλά το νωρίτερο που μπορώ να φτάσω θα είναι 9.30 εάν δεν υπάρχουν προβλήματα στο δρόμο. Δεν μπορώ λοιπόν να υποσχεθώ 100% ότι θα βρίσκομαι εκεί. Λυπάμαι πάρα πολύ έχω και μικρά παιδιά, οπότε μου είναι πολύ δύσκολο να φύγω Κυριακή από τη Σουηδία για να φτάσω στο Στρασβούργο ε, Δευτέρα βράδυ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Ε, μίλησα με τον κύριο Μόντι την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και την Τρίτη και έχουμε ήδη συζητήσει τα θέματα που αναφέρθηκαν και ένας από τους στόχους με τον πίνακα αποτελεσμάτων είναι να, σιγά σιγά να γίνουν ομογενή τα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για το μωρό της ε, πρώην Επιτρόπου Κούντεβα. Δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά με τη μία. Θα πρέπει ε, να αναπτύξουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων ε, στη διάρκεια κάποιων ετών. Η νομοθεσία για τους καταναλωτές στα διάφορα κράτη-μέλη διαφέρει και γι' αυτό ε, υπάρχουν διαφορές στην πρόοδο και γι' αυτό θα απαιτήσει χρόνο το όλο εγχείρημα. Θα πρέπει να είμαστε υπομενετικοί. Θα ήμουν ευγνώμων εάν ο κύριος... Α, έφυγε ο κύριος αυτός. Ε, θα πρέπει να συζητήσω μαζί του στην ε, συνάντηση των σχεδόν ε, ε, εισηγητών. Θα κλείσω εδώ. Ελπίζω να φτάσω εγκαίρως στη συνάντηση στις 8 Φεβρουαρίου, ειδικά αν το θέσετε αυτό ως τελευταίο θέμα στην ημερησία διάταξη μετά τις 9.30 και θα συζητήσω και με τους κοιόδης για πιθανές προσθήκες και συμβιβασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Φοβάμαι ότι δεν θα... Έχουμε χρόνο για την Κομισιόν, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι πολλοί που ακούνε. Θα πρέπει να κλείσουμε πολύ γρήγορα. Ε, ας κλείσουμε εδώ. Θα σας ε, στείλουμε ένα ιδιαίτερα γρήγορο αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο για να σας φέρει στο Κοινοβούλιο. Και θα βάλουμε το θέμα σας τελευταίο στην ημερήσια διάταξη, διότι όπως σας είπα... Ο... Με ενδιαφέρει πολύ να έχουμε πλήρη συζήτηση και θέλω να είναι εκεί όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Εσείς και εγώ και η κυρία Κέπχαρτ. Και Είμαστε εδώ, όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος. Έχουμε κάνει εξαιρετικά πολλή δουλειά τα, τις τελευταίες τέσσερις μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Λήξη της συνεδρίασης και θα τα πούμε στις 8 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.